Καλημέρα σας. Ξεκινώντας θα ήθελα να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους σε αυτή τη μεγάλη ελπίζω συζήτηση για την πολιτική στον τομέα του διαστήματος. Σε δύο τμήματα θα διαρρεθεί αυτή η συζήτηση. Η πρώτη αφορά τη διαστημική πολιτική και την ασφάλεια και γι' αυτό έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Λορέντσικ υπεύθυνο του Δορυφορικού Κέντρου, η κυρία Σιλβέιρα Ράις, της Μονάδας Στρατιωτικών Δυνατοτήτων, τον αντινάβαρχο Τριουλέρ, της Υπηρεσίας Συλλογής Στοιχείων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας του Διαστήματος, του κύριο Αγγούστο Γκονσάλες, του Τμήματος Διαστημικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριος Ντουαμέλ επίσης από την Ευρωπαϊκή υπηρεσία διαστήματος. Το δεύτερο τμήμα θα ασχοληθεί με θέματα ασφάλειας στο διάστημα. Έχει προσκληθεί ο Κρίστιαν Μπέρτ, διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφαλείας, ο κύριος Μάρκο Μαλακάρνα, υπεύθυνο του τμήματος έρευνας. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και θα ήθελα να αφιερώσουμε στη διαστημική πολιτική δύο ώρες και ένα τέταρτο και μία ώρα και ένα τέταρτο στην ασφάλεια και άμυνα. Και έρευνα, συγγνώμη. Θα ακούσουμε πρώτα τις ομιλίες και μετά θα ακούσουμε τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Το ίδιο θα κάνουμε και στη δεύτερη συνάντηση. Για να μην χάσουμε περισσότερο χρόνο, δίνω τον λόγο στον πρώτο ομιλητή. Ξεκινάμε. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μιλήσω στα μέλη της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας για το τι κάνουμε στο δορυφορικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πολύ σημαντικό στα θέματα της ε, παροχής πληροφοριών και υποστήριξης για γεωγραφικές πληροφορίες και τη σχέση του με την ασφάλεια και την άμυνα. Έχω, παρουσια... Έχω προετοιμάσει κάποιες διαφάνειες σχετικά. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε σαφή βασική νομική βάση την κοινή δράση του 2002 που αναφέρει ότι η αποστολή του δορυφορικού κέντρου είναι να στηρίζει τη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα της ε, ΚΕΠΑ ειδικά και μετά της μεταρρύθμισης της ε, συνθήκης της Λισαβόνας ε, παρέχοντας ε, δορυφορική απικό άλλες γεωγραφικές υπηρεσίες. Και επίσης λειτουργούμε και στα πλαίσια της Επιτροπής Πολιτικής Ασφαλείας καθώς και υπό την αιγίδα της υψηλής ε, εκπροσώπου για τις εξωτερικές υποθέσεις ε, της Βαρόνης Άστον, η οποία μας ε, δίνει σημαντικά καθήκοντα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε για τις αναλύσεις μας προέρχονται τόσο από εμπορικές όσο και από κυβερνητικές πηγές. Χρησιμοποιούμε εμπορικές εικόνες δορυφορικές τις οποίες αγοράζουμε στην ελεύθερη αγορά και είναι αλήθεια ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση τα τελευταία χρόνια κάτι μας επιτρέπει να αγοράζουμε δεδομένα υψηλής ανάλυσης που μας επιτρέπουν να κάνουμε τις αναλύσεις μας το διάγραμμα εδώ βλέπετε πώς αυξάνεται τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα των δεδομένων. Επίσης ε, σχεδιάζουμε και νέες ε, αποκτήσεις ε, δεδομένων στο μέλλον που ελπίζουμε ότι επίσης θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Επίσης έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κυβερνητικά δεδομένα. Πριν από ένα χρόνο περίπου εμείς Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Βέλγιο συμφώνησαν να δώσουν πρόσβαση στα στοιχεία του Χέλιος καθώς και στο κόσμο SkyRed, ένα πρόγραμμα ιταλικό για την επαλήθευση δεδομένων. Επίσης διεξάγονται διαπραγματεύσεις για να αποκτήσουμε πρόσβαση και σε ένα άλλο εξαιρετικό κυβερνητικό εργαλείο, το γερμανικό Ζαρ Λούπε. Επίσης έχουμε ξεκινήσει τις πρώτες επαφές για να δούμε αν μπορούμε να αποκτήσουμε και πρόσβαση σε άλλο ένα εργαλείο, το impaired. Η πολιτική μας όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα είναι ότι πρέπει να βασιζόμαστε όσο μπορούμε σε ευρωπαϊκά δεδομένα. Όμως, εφόσον έχουμε και εμπορικές σχέσεις, πρέπει να απλώνουμε τα δίκτυα μας και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούμε κυρίως δεδομένα από τις Ηνωμένε Πολιτείες κυρίως ηλεκτροοπτικά δεδομένα, απεικονίσεις με ραντάρ. Βεβαίως στις απεικονίσεις με ραντάρ βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και σε, στα δεδομένα των ευρωπαϊκών ραντάρ. Το δορυφορικό κέντρο ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση γιατί πρόκειται για πολύ ευαίσθητα δεδομένα και καταλαβαίνουμε λοιπόν πως η εμπιστοσύνη παρασχέθηκε στο δορυφορικό κέντρο. Όσον αφορά τους πελάτες μας τώρα, έχω ακούσει μια εκτίμηση ότι το κέντρο αναπτύχθηκε εξαιτίας της ε, ταχείας ανάπτυξης του ESBD. Και συμφωνώ με αυτό γιατί όντως πρόκειται για μια επιχείρηση πολιτική στρατιωτική που επιτρέπει ολοκληρωμένη ανάπτυξη με δυνατότητες πολιτικές και στρατιωτικές. Στο χάρτη με τις ευρωπαϊκές αποστολές που είναι πληρέστατος βλέπετε ότι υποστηρίζουμε μεγάλη ποικιλία τόσο πολιτικών όσο και στρατιωτικών επιχειρήσεων. Για πέρυσι βλέπετε από άποψη καθηκόντων ότι είμαστε καθαρά πολιτικός οργανισμός αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε συνεργασία και με τις Αμερικανικές στρατιωτικές υπηρεσίες και επίσης πελάτες μας είναι η Αταλάντα όπου υποστηρίζουμε κυρίως πολιτικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα την αποστολή στη Γεωργία ή το Κόσοβο. Είναι αλήθεια όμως ότι το μικρό δυναμικό μας δεν μας έχει επιτρέψει να αναπτυχθούμε πλήρως και παντού. Όσον αφορά το προϋπολογισμό μας, είναι σταθερό στα τελευταία εννέα χρόνια. Παρόλα αυτά, η απόδοσή μας έχει τριπλασιαστεί ή τετραπλασιαστεί αν λάβουμε υπόψη τα έργα που έχουμε αναλάβει. Όμως μέχρι στιγμής ε, δεν έχει υπάρξει συνένεση προκειμένου να αυξηθεί ο προϋπολογισμός μας. Βλέπετε εδώ στο διάγραμμα ότι παρόλο που αυξήθηκαν τα έργα μας από τα 22 το 2002 στα 116 σήμερα έχουν μειωθεί τα καθήκοντα του κεφαλαίου 3. Περνάω σε κάποια παραδείγματα του τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Η ευρωπαϊκή επιχειρήση στο Τσάντ είναι ένας από τους βασικούς μας πελάτες. Επίσης, Προσπαθούμε να κάνουμε γρήγορη χαρτογράφηση συγχωνεύοντας ε, κυβερνητικά και εμπορικά στοιχεία και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αναλυτικά προϊόντα τόσο απόρριτα όσο και όχι, όσο και μη απόρριτα σε ορισμένες περιπτώσεις. Και επίσης αυτή τη στιγμή ο βασικός μας, ο μεγαλύτερος μας πελάτης είναι η ΝΑΦΟΡ στη Σομαλία όπου προσπαθούμε να δώσουμε εικόνες κυρίως όσον αφορά τα, τις θέσεις των πειρατών αλλά και άλλους χερσαίους στόχους. Ανέφερα πλην το Κωσυφοπέδιο και τη Γεωργία που είναι επίσης μεγάλοι πελάτες μας οι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις στο Κωσυφοπαίδιο και την Γεωργία. Άλλα προσεχή παραδείγματα που μπορώ να αναφέρω είναι περιβαλλοντική ασφάλεια, δώσαμε δορυφορικά στοιχεία για την ε, υποβοήθηση των επιχειρήσεων στην IT καθώς και στη Χιλή, τη Μαϊδέιρα και τα λοιπά. Ένα άλλο σημαντικό πρόγραμμα όπου ίσως αναμειχθούμε είναι το πρόγραμμα Space Situation Awareness που αφορά τα αντικείμενα που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη γη Πρόκειται για μια εξειδικευμένη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα του διαστήματος. Τέλος, να πω ότι αναμένουμε με ανυπομονησία την πλήρη εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και την ανάληψη δράσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης καθώς οι περισσότεροι βασικοί μας πελάτες πρόκειται να ενταχθούν σε αυτήν τη νέα αρχιτεκτονική και να λειτουργήσουν με πολιτικού όρους υπό μια κοινή ομπρέλα. Άρα θεωρώ ότι θα αυξηθούν οι απαιτήσει από το δορυφορικό κέντρο. Περνάω στην τελευταία διαφάνεια, προτεραιότητες για το μέλλον. Βελτιστοποίηση των πληροφοριών που διαθέτουμε και συνεχίσα ενημέρωση των κυβερνητικών στοιχείων προκειμένου να βελτιωθεί και η συνεργασία, απλοποίηση της διαδικασίας ανάληψης έργων και αξιολόγηση του δορυφορικού κέντρου μέσω και του GMES. Θεωρούμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της κοινή πολιτικής ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Να πω ότι Πέρυσι είχαμε επισκεφθεί το κέντρο στη Μαδρίτη, μία αντιπροσωπεία μας και εντυπωσιαστήκαμε με το έργο σας αλλά και με το χαμηλό προϋπολογισμό σας. Μας εξέπλησε επίσης το γεγονός ότι δούλευαν άτομα από τόσες πολλές χώρες στο κέντρο σας, ακόμη και ένας Πολωνός. Ευχαριστούμε πολύ τον Διευθυντή. Περνάμε τώρα στην Άλτα Σιλβέιρα Ράισα για το λόγο. Euh, euh, Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Είναι τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα. Προέρχομαι από το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων και Προγραμματισμού. Έχει σαν στόχο τον στρατηγικό ολοκληρωμένο προγραμματισμό για πολιτικές και στρατιωτικές επεμβάσεις της Ένωσης όπως επίσης και το θέμα ανάπτυξης δυνατοτήτων και εταιρικών συνεργασιών. Συντονισμού δηλαδή των διαθεσίμων δυνατοτήτων των κρατών μελών. Ασχολούμεθα επίσης και συνεργαζόμαστε στενά και με το κέντρο δορυφόρων, όπως επίσης και με την πρώτη διεύθυνση της υπηρεσίας της υπάτου εκπροσώπου για τις εξωτερικές σχέσεις. Στα πλαίσια της διαχείρισης κρίσεων μας ενδιαφέρει το θέμα της ασφάλειας. Είναι κάτι το οποίο ανήκει και στη συνθήκη, αλλά είναι και κάτι το οποίο επιτρέπει να εξελιχθεί η γενικότερη στρατηγική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τα δει κανείς αυτά στο διάστημα, είναι αλήθεια ότι το διάστημα θα παίξει ένα ρόλο ο οποίος παραμένει περιθωριακό σε σχέση με άλλες δυνατότητες οι οποίες γίνονται αντιληπτές σαν πλέον επίγοντες, επίγουσες, συγγνώμη, αλλά δεν πάβει ο ρόλος του διαστήματος να είναι βασικός λόγω της μοναδικής ξεχωριστής φύσης του χώρου στο διάστημα. και από το φυσικό περιβάλλον, το οποίο δίνει δυνατότητες προγραμματισμού σε σφαιρικό και στρατηγικό επίπεδο και λόγω του μη, ε, θα έλεγα, παρεμβατικού χαρακτήρα που έχουν άλλες πλατφόρμες παρακολούθησης, αλλά και λόγω του νομικού καθεστώτος που χαρακτηρίζει το διάστημα που θα πρέπει να εξελιχθεί και να προστατευθεί. Δεν μιλάμε μόνο για το διάστημα, αλλά μιλάμε και για κινδύνους, γιατί και το διάστημα δημιουργεί κινδύνους και σε επίπεδο κινδύνων και επίλυσης προβλημάτων θα συνεχίσω την παρουσίασή μου. Θα θέσω δύο ερωτήσεις. Εάν δεν έχουμε στη διάθεσή μας μια διαστημική δεδομένη δυνατότητα, τι θα συμβεί σε επίπεδο κινδύνων. Και αντίθετα, ποιοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι δημιουργούνται από ορισμένα διαστημικά συστήματα στις δραστηριότητες ασφαλείας όπως σε ό,τι μας αφορά η διαχείριση κρίσεων. Σας είπα ότι όλες οι διαστημικές δυνατότητες είναι χρησιμότατες και απαραίτητες για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τη διαχείριση των κρίσεων και είναι μάταιο να προσπαθήσει να επιλέξει κανείς ανάμεσα σε διαφορετικές τέτοιες δραστηριότητες όπως τηλεπικοινωνίες, ναυσιπλοεία, GPS ή ε, το λεγόμενο timing, η χρονοθέτηση. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία που παίζουν ρόλο, ονογραφικά, μετεωρολογικά κτλ. Αν δεν έχουμε αυτές τις δυνατότητες, τότε υπονομεύεται και χειροτερεύει η δυνατότητα ανταπάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμοποιούμε κυρίως τις υποδομές, εμπορικές διαστημικές υποδομές, οι οποίες συμπληρούνται από ορισμένα συστήματα εθνικά κυβερνητικά που τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος του κέντρου. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι δεν έχουμε πάντα τον πλήρη έλεγχο αυτών των υποδομών. θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια πιο συνεκτική απάντηση, η οποία να συμπεριλαμβάνει τα συστήματα ασφαλείας τα οποία είναι διαθέσιμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι, θα πρέπει να υπάρχει, ότι μπορεί να υπάρχει σήμερα μια πλήρως ολοκληρωμένη διαστημική δομή που καλύπτει όλες τις ανάγκες της Ευρώπης σήμερα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο με τους εμπλεκόμενους στον τομέα της ασφάλειας και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ταυτόχρονα το πώς να απαντήσουμε στις ανάγκες τους, το πώς να εντάξουμε στο σύστημα αυτούς τους ιδίους εμπλεκομένους και τα συστήματα τα οποία ελέγχουν, όπως επίσης και ε, τους κυβερνητικούς αλλά και εμπορικούς εταίρους, και να εντάξουμε τα υπόλοιπα διαθέσιμα συστήματα τα οποία χρήζουν ανάπτυξη Να επανέλθουμε λίγο στα θέματα της παρατήρησης του πλανήτη για να σας δώσω ένα παράδειγμα των προβλημάτων και των προκλήσεων. Το δορυφορικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πλέον σωρεύσει μια μακρά εμπειρία στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και κοινή άμυνας έτσι ώστε να μας βοηθήσει και να καταλάβουμε, να λάβουμε αποφάσεις και να ανταποκριθούμε σε καταστάσεις κρίσης. Το κέντρο της Τορεχών έχει στη διάθεσή του αρκετά μέσα, όπως την εμπορική απεικόνηση, τη δορυφορική, αλλά και την δυνατότητα πρόσβαση σε κάποια δορυφορικά μέσα με δεδομένα και εικόνες ε, κυβερνητικά και οπτικά και με ραντάρ έχει επίσης στη διάθεσή του ικανότατους ε, αναλυτές και αυτό είναι μια προστιθέμενη αξία για την ύπατη εκπρόσωπο η οποία έχει πλέον δυνατότητες βελτιωμένες και αυτό είναι χρήσιμο και για το Συμβούλιο και για τη μία. Τώρα, στα πλαίσια του προγράμματος ΖΕΟΕΣ για την προώθηση των συνθήκων ασφαλείας είναι ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα χρήσιμο σε επίπεδο διαστημικό και έχει και χερσαίες βέβαια διαστάσεις. Η πραγματικότητα σήμερα σε επίπεδο αντίληψης της ασφάλειας είναι η εξής αναφέρομαι στη σύνδεση την διοδιευθυντική αν θέλατε ανάμεσα στον παράγοντα ασφαλείας ή έλλειψης ασφαλείας. Ο πολλαπλασιασμός περιβαλλοντικών κρίσεων όπως η Αιτή, η Μαδέρα, η Χιλή κινητοποιούν πολλά μέσα στρατιωτικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν μέσα επιπλέον και επιμέρους στρατιωτικά για πολιτικούς λόγους. Θα βασιστούμε λοιπόν στις ικανότητες τις οποίες ήδη έχουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το Διαστημικό Κέντρο και το ΖΕΟΕΣ είναι μια συνολική απάντηση η οποία λόγω της συνεργασίας η οποία θα το χαρακτηρίζει θα καλύπτει τις ανάγκες μας σε επίπεδο διαστημικής πολιτικής προστατεύοντάς μας από διάφορους κινδύνους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους φόβους τους οποίους εκφράζουν ορισμένοι εμπλεκόμενοι στον τομέα της ασφαλείας οι οποίοι πιστεύουν ότι το ΣΕΡΟΕΣ θα δημιουργήσει προβλήματα στις δικές τους μεθόδους διαχείρισης κρίσεων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους ή εις βάρος τους. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν τους φόβους αυτών των εμπλεκομένων ε, για τον τομέα της ασφαλείας στο διάστημα. Να μιλήσω για τρεις τομείς ε, της ασφάλειας στο διάστημα. Διασφάλιση δεδομένων πρώτο, διασφάλιση των διαστημικών υποδομών δεύτερο και τρίτον το ευρύτερο θέμα της ανεξαρτησίας και της δυνατότητας πρόσβασης στο διάστημα για τις ευρωπαϊκές χώρες. Για το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και επανέρχομαι στο GMS. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να στηριχθεί από το Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων διατηρώντας σεβόμενη μια βασική αρχή που είναι η ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Χαίρομαι λοιπόν εδώ να αναφέρω ότι τον Ιανουάριο η Επιτροπή Ασφαλείας στο διάστημα του Συμβουλίου ε, προτείνει ένα έγγραφο το οποίο αναφέρεται στο σύνολο του ΣΕΡΕΣ και προτείνει λύσεις για τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση του προγράμματος. Θυμίζω ότι η ίδια Επιτροπή Ασφαλείας του Συμβουλίου έχει εμπλακεί ε, στενά και στο πρόγραμμα ε, Γαλιλαίο σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις ασφαλείας. Για τις υποδομές τώρα. Η χρήση του διαστήματος είναι κάτι το πάρα πολύ συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας μια αυξανόμενη εξάρτηση από διαστημικά μέσα. Η εξάρτηση αυτή όμως είναι θα έλεγα αρκετά διάχυτη της φύσης και θα πρέπει εδώ να θέσουμε ένα ερώτημα. Σε ποιο βαθμό έχουμε πράγματι στη διάθεσή μας μια αυτόνομη διάθεση παρατήρησης της γης μέσω των κυβερνητικών ε, ε, δορυφόρων. Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για την αξιοπιστία των δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται και συνδυάζονται. Δηλαδή από τη μία χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες ενός δορυφόρου, από την άλλη όμως δεν είμαστε σίγουροι για τα στοιχεία τα οποία οδηγούν στην σύνθεση αυτών των δυνατοτήτων. Και στόχος λοιπόν του συστήματος ε, της γνώσης των προβλημάτων στο διάστημα είναι κάτι το οποίο ε, θα απασχολήσει τους επόμενους ομιλητές, το Space Situational Awareness. Τώρα, η ανεξαρτησία της υπηρεσίας αυτή. Είναι κρίσιμο θέμα. Τίθεται εδώ το ερώτημα, κάπως προκλητικά αν θέλετε, αν θα πρέπει να θεωρήσουμε τα διαστημικά συστήματα α, κρίσιμες υποδομές. Γιατί η ασφάλεια στο διάστημα είναι προϋπόθεση πολλές φορές για να μπορούν να χρησιμοποιήσουμε μια αρχιτεκτονική διαστημική και για θέματα ασφαλείας αλλά και για άλλες δραστηριότητες. Είναι αλήθεια ότι η ασφάλεια στο διάστημα είναι αν θέλετε μια σφαιρική έννοια η οποία ξεπερνά τις περιορισμένες σφαίρες ενασχόλησης των διαστημικών υπηρεσιών των χωρών. Τίθεται το θέμα λοιπόν των κρίσιμων τεχνολογιών, της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και το θέμα του φάσματος συχνοτήτων που είναι πάντα στα πλαίσια του Γκαλιλαίου υποσυζήτηση. Συμπερασματικά κύριε Αντιπρόεδρε, Έχουμε ένα δεδομένο πλαίσιο για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, αλλά για να μπορέσει η Ευρώπη να αποδείξει ότι είναι μια διαστημική δύναμη, χρειάζεται να αναπτυχθεί και η διάσταση ασφάλεια και διάστημα. Έχουμε ένα θεσμικό μηχανισμό, ξέρουμε πού θα βασιστούμε στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα, στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεπέρασα το χρόνο μου, λέει η κυρία Ράις. Τελειώνω πάντως. Πέρα λοιπόν από τον διαφρομένο διάλογο, νομίζω ότι το, η πρόκληση της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής είναι η ικανότητά της να τεθεί στην υπηρεσία των χρηστών της και στον συγκεκριμένο δικό μας τομέα αναφερόμαστε στους εμπλεκομένους στις διαχειρήσεις κρίσεων. Αυτές είναι οι δύο βασικές προκλήσεις και νομίζω ότι μία μόνο είναι η επιλογή, συνεργασία, συνεργασία και για μια ακόμη φορά συνεργασία. Σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ομιλία και επόμενο είναι ο Ναύαρχος Τριουλέντα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στη σήμερα εδώ προκειμένου να σας ενημερώσω για, την Ευρωπαϊκή, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και να σας μιλήσω για το τι γίνεται στον ε, κοινό χώρο ε, ασφάλειας. Τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με το διάστημα παίζουν σημαντικό ρόλο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Τα καθήκοντά μας στηρίζονται στις συνθήκες και προβλέπουν τέσσερις συνιστώσεις που έχουν να κάνουν άμεσα με το διάστημα. Καταρχάς, να πω ότι θεωρούμε το διάστημα όχι ως δυνατότητα αλλά ως περιβάλλον και ως εργαλείο που βασίζεται σε διάφορα συστήματα. Θα ήθελα τώρα να περάσω σε κάποιες ιδιαιτερότητες των ε, διαστημικών συστημάτων. Καταρχάς, έχουμε έναν χαρακτήρα διτό που μας δίνει πολλές δυνατότητες. Ο οργανισμός μας αφορά κυρίως τις υποδομές, τις δυνατότητες, το δυναμικό. Δυναμικό σημαίνει δημιουργία μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα της άμενας σε διάφορα σε διάφορους χώρους, σε διάφορα θέατρα επιχειρήσεων. Όταν αποφασιστούν τα θέματα τα οποία θα ερευνηθούν, μετά πρέπει να υπάρξει εφαρμογή και εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Επίσης χρειάζεται να γίνεται ενηλογική ανάλυση που αφορά την διακυβέρνηση, την ε, κατάρτιση, το ανθρώπινο δυναμικό κτλ. Ένα πρώτο θέμα που ανέφερα και πριν. Το διάστημα δεν είναι δυναμικό όμως στηρίζει την ανάλυση του δυναμικού και συμμετέχει στην ε, δημιουργία αποτελεσμάτων. Από αυτή την άποψη το διάστημα μαζί με την ε, την έρευνα αναγνώ, την ε, υπηρεσία αναγνώρισης ή το NEC, το Network Capability, βασίζεται κυρίως στους δορυφόρους. Ενώ επίσημα ασχολούν θέματα όπως ε, ο εντοπισμός γεωγραφικής θέσης, η μετεωρολογία και η ωκεαναγραφία. Το διάστημα είναι περιβάλλον. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του από πλευράς αμυντικής. Καταρχάς υπάρχουν κάποιες ζώνες που αναλύονται ιδιαίτερα οι λεγόμενες ε, βάσεις ε, παρατηρήσεων και στις οποίες υπάρχουν πολλά απορρίμματα, υπάρχει μεγάλη συσσόρευση απορριμμάτων και είναι δύσκολη η τοποθέτηση των εργαλείων που χρειαζόμαστε. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό τώρα. Τρίτον, έχουμε ελεύθερη πρόσβαση, όπως είπε και η κυρία Ράις, και επομένως δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη συμπερίληψη. Επίσης, μεγάλη ταχύτητα μετακίνησης, κάτι που βεβαίως είναι δύσκολο εξαιτία των πολλών απορριμμάτων που υπάρχουν στο διάστημα και εξαιτία των θέματων που έχουν να κάνουν με την επιλογή με την επικοινωνία και τις ανταλλαγές. Ένα άλλο θέμα είναι το διαθέσιμο φάσμα. Ας περάσω τώρα στις ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την ασφάλεια. Όπως είπα, το διάστημα είναι ένα περιβάλλον αλλά και ένα σύστημα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας. Χρειαζόμαστε ευελιξία επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε, χρειαζόμαστε να, τρόπους να μπορούμε να συλλέγουμε τις πληροφορίες. Επίσης, πολλές φορές έχουμε έντονη συγκεκριμένη χωρική τοποθέτηση. Βεβαίως ε, η συσχέτιση χερσαίας και διαστημικής διάστασης μερικές φορές είναι εύκολη. Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές απειλές ε, που αντιμετωπίζουμε στο διάστημα. Για παράδειγμα τα απορρίμματα ενώ πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος ε, επιθέσεων. Καταλαβαίνετε επίσης ότι υπάρχουν πολλά συστήματα με ισοδύναμα αποτελέσματα. Και βεβαίως χρειαζόμαστε συνεργασία από την βιομηχανία και ευελιξία, προκειμένου να δημιουργήσουμε εργαλεία με βάση το οικονομικό πλαίσιο που έχουμε στη διάθεσή μας. Τα διαστημικά συστήματα συνεισφέρουν και για πολιτικούς και στρατηγικούς λόγους. Διτό σύστημα λοιπόν. Κάτι που έχει τονιστεί αρκετές φορές και βεβαίως εξαρτώμαστε και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα διαστημικά προγράμματα διακρίνονταν είτε σε πολιτικά είτε σε στρατιωτικά. Αυτό όμω αλλάζει σιγά σιγά για δύο λόγου. Πρώτον, οικονομικοί περιορισμοί. Νομίζω προφανές. Αλλά και οι ανάγκες που εκφράζουν πλέον οι περισσότεροι χρήστες και πολιτικοί και στρατιωτικοί όσον αφορά τις ανάγκες τους για εικόνες, τηλεπικοινωνίες κτλ. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε το δυναμικό προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες τις συλλογικές. Κάθε πρόγραμμα λοιπόν πρέπει να βασίζεται σε έναν οδηγό που θα δείχνει τις ανάγκες, το what for του πελάτη. Είναι λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε συνοηθεί εκ των προτέρων και να μοιραζόμαστε τους ίδιους στόχους. Όταν ο εμπορικός κόσμος μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες, αυτό μας δίνει πολλές δυνατότητες να βρούμε λύσεις και για την ε, ασφάλεια και την άμυνα. Αν και αυτό δεν είναι πάντα δυνατό στην περίπτωσή μας. Όμως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες προϋποθέσεις όπως η προστασία των δεδομένων. GMES και το δεύτερο πρόγραμμα, έχουμε δηλαδή δύο προγράμματα που έχουν να κάνουν με το διάστημα, ένα πολιτικό και ένα στρατιωτικό. Πρέπει να εξετάσουμε τις ενέργειες που μπορούν να προκύψουν. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουμε κάθε φορά εκ των προτέρων και αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ήδη ξεκινούν να το καταλαβαίνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι άλλοι φορείς. Έχουμε κοινέ δράσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανήμινας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έχουμε καθαρά στρατιωτικά θέματα όπου δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ένα Τελευταίο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή στηρίζουμε ένα πρόγραμμα TASK που έχει να κάνει με την επικοινωνία μέσω δορυφόρου και θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μάλι να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας με την καλύτερη δυνατή τιμή. Περνάω τώρα σε κάποιους άξονες που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε στο μέλλον για να έχουμε καλύτερες συνέργειες. Είναι πολλοί οι τομεί στου οποίου μπορούν να υπάρξουν συνεργασίε, αλλά θα πρέπει να είναι και διατρική. Η πρώτη πρόταση είναι να αντικαταστήσουμε την αντίληψη συνολικά για το διάστημα ε, με μία αντίστοιχη η οποία βάζει το διάστημα σε ένα πλαίσιο που να περιλαμβάνει και χερσαίες και διαστημικές εφαρμογές σε ένα σύστημα το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουμε σε επίπεδο δυνατοτήτων. Στόχος είναι να ξεκινήσουμε νωρίς ε, περιγράφοντας την ανάγκη η οποία υπάρχει και στον τομέα τον πολιτικό και στον τομέα τον στρατιωτικό και να ξεκαθαρίσουμε τον χώρο χωρίς να υπάρχουν συγχύσεις ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες, ε, σχεδιάζοντας τα προγράμματα ε, και τα στρατηγικά και τα ερευνητικά και αναπτυξιακά. Να φέρουμε σε επαφή το στρατιωτικό με τον πολιτικό τομέα για να συστηματοποιήσουμε περισσότερο τις διαθέσιμες συνέργειες. Σας ευχαριστούμε και η επόμενη ομιλητρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Βίμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη γιατί αντικαθιστώ τον κύριο Αυγούστο Γκοντζάλες, ο οποίος είναι επικεφαλής της Μονάδας Συστημικής Πολιτικής και Συντονισμούς. Ε, βρίσκεται σε μια συνεδρίαση με τον Επίτροπο Ταγιάννη, λοιπόν. Πρωτού ξεκινήσω να εξηγώ τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα του διαστήματος και της ασφάλειας να εξηγήσω πού εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον τομέα της πολιτικής αυτός. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για το Διάστημα που καταρτίστηκε το 2007 τονίζει ποια μπορεί να είναι η συμβολή του διαστήματος ε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της Ένωσης ε, από όλες τις προκλήσεις που μπορεί να επηρεάσουν τους Ευρωπαίους πολίτες καθώς και τις ε, συμπεριλαμβανομένων μάλλον και των στρατιωτικών προκλήσεων. Η πολιτική αυτή δημιουργεί τη σχέση μεταξύ της διαστημικής διάστασης και του ESDP με μια, ένα συνδυασμό στοχιωτικών και μη ε, λύσεων. Η ευρωπαϊκή πολιτική για το διάστημα αναγνωρίζει επίση ότι οι τεχνολογίε για το διάστημα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για πολιτικούς και για στρατιωτικούς σκοπού για να βελτιωθεί ο συντονισμό μεταξύ αμυντικών προγραμμάτων και πολιτικών προγραμμάτων, λαμβάνοντα υπόψη τι απαιτήσει και των δύο τομέων, των διαφορετικών αρμοδιοτήτων και το 2008 το Συμβούλιο για το ψήφισμα του Συμβουλίου για το διάστημα έλαβε και συμπεριέλαβε την ασφάλεια μεταξύ των τεσσάρων προτεραιοτήτων για την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής αυτής για το διάστημα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του το 2008 τονίζει τη σημασία της πολιτικής για το διάστημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας το διάστημα καθίσταται αυτοδύναμη ευρωπαϊκή πολιτική και θα επανέλθω σε αυτό στο τέλος της ε, παρουσίασής μου. Και ο Επίτροπος, ο Πρόεδρος, συγγνώμη παρόσω. ανέφερε το διάστημα ως ε, μία από τις βασικές πέντε προκλήσεις για την επόμενη θετία της Επιτροπής. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, που βρισκόμαστε. Το ψήφισμα του Συμβουλίου του 2008, στο οποίο ήδη αναφέρθηκα, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους σχετικούς φορείς, την Επιτροπή από κοινού το Συμβούλιο, να ιδρύσουν ε, έναν ε, δομημένο διάλογο για την ασφάλεια και τι το διάστημα με σκοπό να εφαρμοστούν τα όσα έχουν αναφερθεί θεωρητικά. Να εξεταστούν δηλαδή πρακτικοί τρόποι συνεργασιών μεταξύ πολιτικών ε, σκοπών, δραστηριοτήτων και στρατιωτικών δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά το διάστημα προκειμένου να συμβάλλει η διαστημική πολιτική στις ε, δραστηριότητες ασφάλειας και στον τομέα τον πολιτικό και στον τομέα το στρατιωτικό. Και αυτός ο δομημένος διάλογος ε, ε, αναφέρεται στην Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την ΙΖΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους θεσμικούς φορείς. Άρα, για μας, θεσμικό επίπεδο, πρόκειται για το πρώτο μέσο με το οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε και να συντονίσουμε καλύτερα τις δραστηριότητές μας. Επιπλέον, και το ανέφεραν άλλωστε και οι προηγούμενοι ομιλητές, έχουμε το GMS. E σε ό,τι αφορά τη χρήση του GMS e στον τομέα της ασφάλειας. Η ναυτική, η παρακολούθηση των συνόρων, η παρακολούθηση της ναυτικής περιοχής έχουν εντοπιστεί ως ε, προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια και αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει σε επίπεδο επιτροπής καταρχάς να δούμε ποιες είναι οι απαιτήσει χρήστη. Να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες των διαφόρων χρηστών που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές GMES σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Και να τονίσουμε και αυτούς τους τρεις ε, τομείς που ανέφερα. Για να προχωρήσει η συνιστόσα της ασφάλειας σε ό,τι αφορά το GMES, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντοπίσει ποιες είναι οι πληροφορίες οι οποίες ε, αφορούν τον τομέα της ασφάλειας από το GMES και πώς ε, οι τομείς αυτής μπορούν να ενισχύσουν, για παράδειγμα, τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες. και πού οι εφαρμογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ασφάλειας. Να εντοπίσει επίσης κατά πόσο χρειαζόμαστε περισσότερα, κατά πόσο χρειαζόμαστε επιπρόσθετες ε, υπηρεσίες ε, ασφάλειας, επιπρόσθετες δυνατότητες, ικανότητες σε ό,τι αφορά τα GMES, το GMS. E επίσης, εξετάζουμε πώς ε, τα κράτη-μέλη και πώς οι στρατιωτικές ε, ανάγκες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του GMS, Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας έχει δώσει εντολή εξέτασης ε, σχετικών απαιτήσεων και έχουν γίνει σχετικές εκκλήσεις και αποψηφίσματα του Κοινοβουλίου. Τέλος, για, για τις στα κριτικό σκέλος και τις κριτικές ανάγκες μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας, τα στοιχεία είναι ακόμη συζήτηση. Να έχουμε επίσης υπόψη ότι υπάρχει έντονη συνεργασία και είναι απαραίτητη αυτή με τους ε, εμπλεκόμενους φορείς από όλη την κοινωνία και επίσης προσπαθούμε να αποφύγουμε αλληλεπικάλυψη. Κατά δεύτερον, έχουμε το Γαλιλαίο Αναφέρεται ότι τα συστήματα αυτά, ενώ μεν σέβονται τον πολιτικό τους χαρακτήρα, ενδεχομένως τέτοια συστήματα να έχουν και στρατιωτικές χρήσεις, και θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς ε, και με ποιο τρόπο τα πρόγραμμα Γαλιλαίος θα μπορούσε να παράσχει υπηρεσίες ως προς την ασφάλεια. Έχουμε μαζί μας εδώ στην αίθουσα δύο συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις υπηρεσίες για το Γαλλιέλεο, που εντάσσεται στη γενική μας διεύθυνση. Άρα, αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις για το Γαλιλαίο, ε, ευχαρίστως να σας απαντήσουν οι συνάδελφοι για το που βρισκόμαστε σήμερα. Και κατά τρίτον, πέρα από τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το πώς χρησιμοποιείται το διάστημα για την ασφάλεια επί της γης, έχουμε άλλη μια διάσταση της ασφάλειας και του διαστήματος, το πώς θα διασφαλίζεται η ασφάλεια των, ε, του διαστήματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού την ΙΣΑ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία δραστηριοποίησης και ευαισθητοποίησης για το διάστημα. Θα ακούσουμε μάλλον ε, διάφορες πληροφορίες για την ε, προπαρασκευαστική διαδικασία που ξεκίνησε η ΙΖΑ πέρυσι και το ψήφισμα του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για το διάστημα θα ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, πρέπει να παίξει ε, σημαντικό ρόλο για την ε, διαχείριση ενός μελλοντικού τέτοιου συστήματος και επίσης ε, απευθύνθηκε και ανέφερε για το θέμα και της πολιτικής δεδομένων. βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαλόγου επ' αυτού, περιλαμβανομένη τη ε, ΙΖΑ, του, Γραμματέία του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΝΤΑ, καθώς και των κρατών μελών που παρέχουν σχετικά κονδύλια για την ανάπτυξη μιας ε, μελλοντικής ε, πολιτικής ευρωπαϊκής SSA για την ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Η εκτέλεση, η εφαρμογή τώρα τέτοιων μελλοντικών ε, συστημάτων ε, ευρωπαϊκού SSA ασφαλώς θα αποτελέσει μια πρόκληση για το παρόν οικοδόμημα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και το διάστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για συστήματα εξ αρχής διτής χρήσης και καταλαβαίνουμε φυσικά, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό ενδεχομένως να, ζητήσει, να απαιτήσει νέα συστήματα ε, συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων πυλώνων. Είχαμε μια σχετική συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα στο Μαδρίτη για το TMS e και την SSA έγιναν κάποιες, ε, διατυπώθηκαν κάποιες απόψεις για τη δυτή αυτή χρήση των προγραμμάτων αυτών και το εργαστήριο αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω διαδικασίες για την ασφάλεια και την άμυνα υπό την Βελγική Προεδρία. Τέλος, να πω δύο λόγια για τη Λισαβόνα, τη συνθήκη της Λισαβόνας το άρθρο 189 με το οποίο πλέον το διάστημα και η σχετική πολιτική κατοχυρώνεται ως κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταρτήσει μια ευρωπαϊκή πολιτική για το διάστημα και ότι θα εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα τα οποία ενδεχομένως να διαμορφωθούν ως πρόγραμμα ευρωπαϊκό για το διάστημα για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Τι σκοπεύουμε λοιπόν να κάνουμε, τι σκοπεύουμε να κάνουμε για το άρθρο 189. Βρισκόμαστε σε φάση κατάρτισης μιας ανακοίνωσης για την μελλοντική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, στον τομέα του διαστήματος, όπου θα εντοπιστούν οι βασικές προτεραιότητες τις οποίες σκοπεύει να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επόμενο διάστημα. Η ανακοίνωση θα εκδοθεί το Σεπτέμβριο του 2010 συνειδητοποιούμε ασφαλώς ότι από τη στιγμή που θα ορίσουμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό θα έχει αντίκτυπο κατά μεγάλο βαθμό στις ε, δράσεις τις οποίες αποσκοπεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το διάστημα και την ασφάλεια στο επόμενο διάστημα και θα πρέπει ασφαλώς να ακολουθήσει η νομοθετική διαδικασία για το μελλοντικό διαστημικό πρόγραμμα υπό το πλαίσιο των επόμενων ε, δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020 και η νομοθετική αυτή πρόταση θα κατατεθεί καταρχάς Απρίλιο-Μάιο του 2011. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κλείσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να περάσουμε κατευθείαν στο διάστημα. Στο Ευρωπαϊκό Διάστημα και την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Ο κύριος Ντουαμέλ έχει το λόγο. Προέρχομαι από την ΕΣΑ, την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Δεν είναι υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι διεθνής οργάνωση. Και δύο από τα μέλη μας, η Νορβηγία και η Ελβετία, δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εργαζόμαστε στο διαστημικό χώρο εδώ και 30 χρόνια δημιουργηθήκαμε σαν μια οργάνωση έρευνας και ανάπτυξης. Δεν έχουμε εμπορικέ φιλοδοξίες για την εκμετάλλευση ουδήποτε συστήματος. Όπως είδε, είπε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μια συμφωνία πλαίσιο από το 2004. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας ε, ε, δημιουργούμε και το Συμβούλιο Διαστήματος, ένα Υπουργικό Συμβούλιο δηλαδή των μελών, το οποίο έχει συνεδριάσει μέχρι τώρα έξι φορές κατά τη διάρκεια της τέταρτης συνάντησης του Διαστημικού Συμβουλίου το 2007 υιοθετήθηκε η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική. Ένα από τα βασικά σημεία της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής είναι ότι οι Υπουργοί μας ζήτησαν να καλύψουμε τις ανάγκες της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Συνεπώς όχι μόνο μπορούμε να παρεμβαίνουμε στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, αλλά οφείλουμε να το κάνουμε. Υπάρχουν δύο βασικά προγράμματα τα οποία αναπτύσσουμε στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία στον τομέα της ασφάλειας, καταρχάς το GMES, το οποίο αναπτύσσουμε παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το περιβάλλον και την ασφάλεια και δεύτερον το πρόγραμμα Γκαλιλαίο, το οποίο γνωρίζετε ίσως και καλύτερα από μένα. Ένα πρόγραμμα αναυσιπλοείας. Αναπτύσσουμε και άλλα πολιτικά προγράμματα, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα και για τους στρατιωτικούς χρήστες. Καταρχάς τα συστήματα μεταφοράς δεδομένων που είναι τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Ένα από τα βασικά μέσα το οποίο οποιοδήποτε εμπλεκόμενο στον τομέα έχει ανάγκη είναι η επικοινωνία. Πώς εμείς αναπτύσσουμε ένα στερισμό ε, δορυφόρων που είναι διασυνδεδεμένοι έτσι ώστε οσδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να συνδεθεί με οποιονδήποτε άλλον. Διαστημικά συστήματα όπως συστήματα ε, παρατήρησης της γης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς τα συστήματα μετάδοσης που έχουμε αναπτύξει έτσι ώστε σε πραγματικό χρόνο να βλέπουμε τι συμβαίνει στη γη. Για να σας δώσουμε μια ιδέα του τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Όλα αυτά ελέγχονται φυσικά από τις επίγειες μονάδες, θα πρέπει το σήμα δηλαδή να σταλεί, να ζητηθεί μια συγκεκριμένη αποστολή, ο δορυφόρος πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάρει τις φωτογραφίες, παίρνει τις φωτογραφίες, και θα πρέπει οι φωτογραφίες να έρθουν πίσω στο, ε, στην επίγεια μονάδα για να αναλυθούν. Και με τα δεδομένα αυτά λοιπόν μπορούμε να ζητήσουμε επακριβέστερες αποστολές από τους ε, δορυφόρους στο μέλλον. Το σύστημα αυτό δεν σχεδιάστηκε μόνο για τους δορυφόρους, αλλά χρησιμοποιείται επίσης και ε, για άλλες επίγειες μονάδες, αυτοκινούμενες κτλ. Έχετε ακούσει ήδη ότι η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ξεκίνησε ένα από τα προγράμματα α, χωροθέτησης στο διάστημα. Είναι μια ανάγκη της ίδιας της υπηρεσίας μας, η οποία χρησιμοποιεί πολλούς επιστημονικούς δορυφόρους και είμαστε εξαρτημένοι από τη ΣΥΠΑ, έτσι ώστε να προειδοποιούμεθα αν κάποιοι από τους δορυφόροι μας μπορούν να χτυπήσουν ας πούμε με ε, άλλα τμήματα εγκαταλελειμμένα δορυφόρων κτλ. Έχουμε και ένα άλλο μικρό πρόγραμμα στο οποίο βρισκόμαστε σε μια πρώτη φάση που έχει γίνει δεκτή από τους υπουργούς. Θα δημιουργήσουμε ένα διαστημικό κατάλογο, μια απαρίθμηση δηλαδή του τι κυκλοφορεί γύρω από τη γη, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τυφλά οι δορυφόροι μας. Το δεύτερο είναι ένα επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο ε, δίνει λειτουργικές υπηρεσίες όταν εκτοξεύεται ύλη από τον ήλιο προς τη γη αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ε, καταστάσεις και στο διάστημα Θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να προειδοποιεί τις περιοχές οι οποίες έχουν ε, ε, ευαίσθητα συστήματα, όχι μόνο διαστημικά, αν υπάρχει πρόβλημα με τις ε, ηλιακές εκρήξεις για να προστατευθούν από το φαινόμενο. Ένα τρίτο τμήμα είναι το Near Earth Object. Προσπαθούμε ουσιαστικά να ανοιχνεύουμε τα τμήματα βράχων τα οποία πετούν προς τη γη ή κοντά στη γη. Ε, μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα και δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιου είδους καταστροφές όπως αυτή που ε, συνάντησαν οι ε, δεινόσαυροι κάποτε στη γη. από το 1998 αριθμός των αντικειμένων που έχουμε ανοιχνεύσει να έρχονται προς τη γη έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη επιστημονική αντίληψη του τι ακριβώς συμβαίνει. Και το τελευταίο τμήμα είναι η διαδικτύωση και το κέντρο δεδομένων. Η διαστημική υπηρεσία δεν έχει, δεν έχει σαν εντολή το να μελετά τη διακυβέρνηση τέτοιου είδους συστημάτων. Εδώ συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει γιατί δεν αρκούν ε, τα τηλεσκόπια για να δούμε τι πλέει στο διάστημα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι ε, εμπιστευτικά και χρειάζεται μια συνολική αντιμετώπιση του προγράμματος αυτού. Αυτό το οποίο είναι σε ενέργεια σε αυτή τη φάση είναι η χάρτα για τις καταστροφές. Η χάρτα αυτή για τις καταστροφές δημιουργήθηκε από την Γαλλική Διαστημική Υπηρεσία εδώ και 10 χρόνια Έχουμε υποσχεθεί σε όλους όσους έχουν αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές στη χώρα τους να τους δίνουμε δωρεάν διαστημικά προϊόντα. Οι χώρες και οι οργανώσεις οι οποίες ε, συνδέονται με την χάρτα αυτή ενημερώνονται δωρεάν στις αρχικές φάσεις ε, για τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ενεργοποίηση σε εβδομαδιαία βάση αυτής της χάρτας να σας δώσω κάποια παραδείγματα από πράγματα που έχουμε κάνει. Ένας κυκλώνα στον Ειρηνικό ωκεανό τον μήνα Φεβρουάριο σαν παράδειγμα. Δεν ήταν μείζον θέμα στις ειδήσει στην Ευρώπη, όλα αυτά υπήρξαν ε, πολλά προβλήματα για τους Ευρωπαίους τουρίστες που ήταν εκεί και δώσαμε τα απαιτούμενα στοιχεία. Οργανώσαμε στο παρελθόν και πολλές διασκέψεις και συναντήσεις με τις κοινότητες των Χριστών ε, συγκεντρώνοντας την προσοχή μας στους πολιτικούς χρήστες. Έχουμε επίσης συνεργαστεί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Έχουμε οργανώσει το Φόρουμ Καινοτομία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και είμαστε σε συνεχή επαφή και με άλλους που ασχολούνται με τα ίδια θέματα στην Ευρώπη. Εδώ είναι κάποιες από τις ανάγκες και τα κριτήρια που έχουν οι χρήστες μας. Έχουμε εντοπίσει τέσσερα βασικά θέματα τα οποία θέλουν οι χρήστες μας ε, να μας απασχολήσουν και ακούστηκαν στις ε, παρουσιάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών. Υπάρχει πρώτον μια πραγματική ανάγκη για μια εγγυημένη πρόσβαση σε δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα περισσότερα δεδομένα προέρχονται από εμπορικούς χρήστες και μη ευρωπαίους εμπορικούς χρήστες. Η Ευρώπη εξαρτάται εν πολλής από εμπορικούς παροχής στοιχείων. Δεν είναι βέβαια, δεν είναι ε, σίγουρα τα πράγματα, δεν είναι δεδομένο το ότι θα έχουμε τα στοιχεία που θέλουμε όταν τα θέλουμε. Είναι επίσης και εμπορικό το πρόβλημα, δίνουμε πάρα πολλά χρήματα σε αυτούς τους μη ευρωπαίους εμπορικούς ε, δορυφόρους, γιατί να μην τα δίνουμε σε ευρωπαϊκούς δορυφόρους. Το GMES, ξέρετε ε, ε, τι είναι, είναι προγράμματα τα οποία αντιμετωπίζονται ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Αυτό μερικές φορές δημιουργεί προβλήματα, θα πρέπει να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση των προγραμμάτων αυτών έτσι ώστε να βλέπουμε τα διαστημικά συστήματα σαν ένα ενιαίο σύστημα την παρατήρηση του πλανήτη, δηλαδή την, τις τηλεπικοινωνίες, τις επικοινωνίες γενικότερα και την αυσιπλοεία, ε, να τα αντιμετωπίσουμε όλα ε, ενιαία και ολιστικά. Αυτό θα μειώσει και το κόστος. Ε, θα πρέπει να καλύψουμε επίσης και τη διάσταση των χερσαίων τηλεπικοινωνιών που πολλές φορές εξαρτώνται από τις διαστημικές υπηρεσίες Πρέπει να βελτιώσουμε τις δυνατότητες που έχουν τα δίκτυα στο μέλλον. Υπάρχει επίσης ε, αίτημα να είμαστε πιο γρήγοροι στις απαντήσεις μας. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε τα δεδομένα διαθέσιμα νωρίτερα. Μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα του τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Έχει αποδειχνεί ότι αν η Ευρώπη πρέπει να παίξει το ρόλο ενός σφαιρικού παράγοντα, δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από άλλους, αλλά πολλές φορές περιμένει και τους άλλους χρήστες. Αν περιμένεις να πάρεις στοιχεία από άλλους χρήστες δεν έχεις καμία προτεραιότητα και πρέπει να περιμένεις πριν σου δώσουν τις πληροφορίες που χρειάζεται. Θέλουμε επίσης να δίνουμε τα προϊόντα αυτά σε αυτούς οι οποίοι τις έχουν ανάγκες και αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν στρατηγικής φύσης αποφάσεις. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και ποιες είναι οι τεχνολογίες με τις οποίες κάτι τέτοιο θα γίνει εφικτό. Και τέταρτο θέμα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει είναι ότι πολλοί ε, θεωρούν ότι η διαστημική πολιτική είναι ένα πλεονέκτημα και πρέπει να καλύψουμε έτσι τις ε, ανάγκες οι οποίες υπάρχουν σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει η διαστημική αυτή παρέμβαση. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει σαν Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία να δούμε με ποιο σφαιρικό τρόπο αντιμετωπίζουμε τα θέματα της ασφάλειας και άμυνας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα μητρικό, ένα σύστημα συστημάτων για τηλεπικοινωνίες, για αναυσιπλοεία, βασιζόμενοι στην αρχή της επικουρικότητας. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον υπάρχουν εθνικά στοιχεία πρέπει να τα συνδυάσουμε με το σύστημα για να γίνει όσο πιο αποδοτικό γίνεται και να ικανοποιήσει όσους περισσότερους χρήστες γίνεται. Το σύστημα αυτό έχει χαρακτηριστεί χρήσιμο κυρίως για χρήση πολιτικών υπηρεσιών στον τομέα των κρίσεων. Δεν εξαιρούμε και δεν αποκλείουμε τους στρατιωτικούς. Πολλές φορές οι στρατιωτικοί εμπλέκονται στη διαχείριση έτσι και αλλιώς των χρήσεων. Το σύστημα παρέχει υπηρεσίες σε όλες τις κοινότητες χρηστών, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δεδομένη η έκφραση των αναγκών του πολιτικού τομέα και πρέπει να καλυφθούν. Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία συνεργάζεται και με τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους Υπουργούς Έρευνας, καλύπτοντας τις πολιτικές ανάγκες κυρίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε στις στρατιωτικές ανάγκες αλλά βασικοί πελάτες μας εισαγωγικά είναι πολιτικοί χρήστες. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Τιουαμέλ. Ευχαριστούμε και όλους τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα τα πάντα. Αυτός όμως είναι ένας καλός λόγος για να σας ρωτήσουμε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και να ακούσουμε κάποιες ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Ε, θα ξεκινήσω εγώ τις ερωτήσεις. Από την επίσκεψή μας πέρυσι στο δορυφορικό κέντρο μας είπατε ότι είχατε πολύ στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι πολλά από τα δεδομένα που χρησιμοποιείται προέρχονται από τους ε, Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και εσάς κύριε Λοβερένσης ε, αλλά και τους δύο οργανισμούς ε, ποια είναι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και άλλες τρίτες χώρες, Ρωσία, Κίνα. Πώς ακριβώς πραγματοποιείται, ποια είναι η εικόνα αυτής της συνεργασίας. Να ακούσουμε πρώτα πέντε ερωτήσεις και μετά τις αντίστοιχες απαντήσεις. Οπότε, αν κάποιος ευρωβουλευτής έχει ερώτηση, παρακαλώ να την κάνει και να μας πει προς ποιον εμπειρογνώμονα απευθύνεται. Κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μερικές ερωτήσεις να θέσω στους ε, ομιλητές. Να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο και στην τελευταία θητεία απασχόλησε το Κοινοβούλιο, όχι μόνο εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών εξετάσαμε τα θέματα ιδιωτικών επενδύσεων για το Γαλιλαίο και την αποτυχία τους και αναλήφθηκαν κάποιες πτυχές από τον προπολογισμό και στην ε, τρέχουσα αυτή δημοσιονομική περίοδο για το, μέχρι το 2013 έχει οριστεί ένα ανώτατο όριο και τώρα ακούμε ότι ενδεχομένως και κατά πάσα πιθανότητα να μην αρκέσει το ποσό αυτό και αναφέρατε κυρία Βίμπνερ ότι θα μπορούσατε να αναφέρετε να πείτε δύο λόγια για το θέμα αυτό σχετικά με το πότε μπορούμε να υπολογίζουμε ότι θα καταστεί λειτουργικό το πρόγραμμα Γαλιλαίος. Αυτό είναι η πρώτη μου ερώτηση. Στην πολιτική μας για το διάστημα, θέλαμε να τονίσουμε, ένα στόχος ήταν να τονίσουμε την ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών τεχνολογιών. Πώς έχει λοιπόν η συνεργασία και ο προγραμματισμός γιατί υπήρχε το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Εκτόξευσης και θα ήθελα να ξέρω πώς έχει, το, πώς έχει η εξάρτησή μας από τη Ρωσία και τους σχετικούς πυράβλους σήμερα. Να μου πείτε επίσης σε ό,τι αφορά το δορυφορικό κέντρο, το EUSE, είδαμε ότι οι απαιτήσει είναι υψηλές και θα πρέπει έχουν ήδη αυξηθεί οι αρμοδιότητες. Το 2008 διπλασιάστηκαν οι αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι παίζουν τον βασικό ρόλο σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για το, την ευαισθητοποίηση και το διάστημα. Οι πόροι αρκούν για την ε, ικανοποιητική εκτέλεση των ε, καθηκόντων αυτών ή μήπως ε, υπερφορτώνεται η υπηρεσία αυτή και δεν έχει τη δυνατότητα με τους πόρους που διαθέτει να εκτελέσει τα καθήκοντα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Η κυρία Γκόμες από τους Σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς επιτρέψτε μου να πω ότι λυπάμαι που δεν μπόρεσα να έρθω εδώ από την αρχή γιατί είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κυρίου Παπανδρέου και ήταν σημαντικό να ακούσουμε τι είχε να πει και εμείς ως εκπρόσωποι των PIGS. Να πω ότι χαίρομαι για το ρόλο που είχε παίξει το Κοινοβούλιο στην εξέβρεση λύσης για τον Καλλιέο πριν από δύο χρόνια. Και να πω ότι τότε θεωρούσαμε ότι οι στρατιωτικές χρήσεις του Γκαλιλαίο, που είναι προφανές όπως είπαν και οι ομελητές μας, θα ήταν όντως χρήσιμες Τότε δεν είχε φανεί αυτό, ίσως γιατί είχαμε διαφορετικά ενδιαφέροντα. Όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και ρωτάω, δεν θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για όλους αν θεωρούσαμε δεδομένες αυτές τις στρατιωτικές χρήσεις του Καλλιλέου. Το δεύτερο ερώτημά μου. Οι Ηνωμένε Πολιτείες υπό την κυβέρνηση Bush δεν είχαν δηλώσει σαφώς, αλλά στην πράξη είχαν εφαρμόσει μια εξαιρετικά επιθετική διαστημική πολιτική που διακήρυσε την ε, κυριαρχία με προγράμματα όπως αυτά της ε, της ε, καταδίωξης των πυρηνικών κτλ. Με την κυβέρνηση Ομπάμα υπάρχει κάποια αλλαγή στην προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης μπορείτε να μας πείτε προς τα που βλέπετε να κατευθύνεται η Κίνα. Αυτό σχετίζεται και με το ερώτημα που ήδη έκανε ο Πρόεδρός μας. Επίσης, ε, την τελευταία φορά που είχαμε συζητήσει το θέμα, κατά την έγκριση της έκθεσης το 2008, είχαμε πει ότι η συνθήκη για το εξώτερο διάστημα χρειαζόταν ε, ενημέρωση και ενίσχυση ειδικά εξαιτίας των προβλημάτων που προκύπτουν από την αύξηση των ε, απορριμμάτων ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει κάποια σχετική δράση. Και τέλος, τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας νομίζω αναγνωρίσαμε ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή οντότητα που θα μπορεί να συντονίζει τις δραστηριότητες σε θέματα ασφάλειας στο διάστημα και η οποία θα διασφαλίζει και την ε, καλή συνεργασία πολιτικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων. Βεβαίως ακούμε ότι εκεί εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες και διάφορα υπουργεία, μεταξύ των οποίων και τα οικονομικά υπουργεία. Τώρα όμως έχουμε την συνθήκη της Λισαβόνας και υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη οντότητα που θα μπορούσε να βοηθήσει στο συντονισμό. Ποια θα είναι η σχέση σας με την είπατε εκπρόσωπο για την εξωτερική δράση. η νέα υπηρεσία εξωτερικής δράσης τι ρόλο θα παίξει στα πλαίσια της παγκόσμιας δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος να πω ότι είχα εντυπωσιαστεί όταν διαπίστωσα τότε με το τσουνάμι στο Άτσε ότι η ευρωπαϊκή τεχνολογία η ευρωπαϊκή δορυφορική τεχνολογία βοήθησε τις αρχές του Άτσε να ταιριάξουν τις δορυφορικές φωτογραφίες πριν και μετά και να μπορέσουν έτσι να δώσουν άδειε στους πολίτες για να ανοικοδομήσουν τα κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Ευχαριστώ πολύ. Από την ΚΟΕ, κύριε ε, κυρία Λούζινγκ, θα ήθελα μετά την κυρία Γκόμα και μετά τον κύριο Γκάλερ να συμφωνήσω και εγώ και να ρωτήσω το εξή. Μα παρουσιάσατε με διάφορου τρόπου ε, τι θα κάνουμε στο άμεσο μέλλον με τις τεχνολογίες αυτές ε, που μας παρουσιάσατε ποιοι είναι οι διάφοροι αυτοί τεράστιοι τομείς οι οποίοι μπορούν να συνδυαστούν και κατέστη ε, σαφές ότι υπάρχει μια έντονη εμπορική διάσταση στο όλο θέμα και φυσικά ότι υπάρχει και μια έντονη διάσταση σε ό,τι αφορά το κόστος. Το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο ε, χρηματοδοτείται από ένα κράτος, ε, από τα κράτη-μέλη, ενώ το GMES ε, χρηματοδοτείται από την κοινότητα. Θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το συνολικό κόστος για το Γαλιλαίο και για το GMS. Ποια είναι η τρέχουσα εκτίμηση επακριβώς. Και θα ήθελα να ξέρω τι ποσοστό χρηματοδοτείται από τον κοινωτικό προϋπολογισμό και κυρίως από ποια κονδύλια. Η κυρία Γκόμες ε, το ανέφερε και εγώ το ίδιο κατάλαβα ότι επιθυμείται η στρατιωτική πτυχή του Γαλιλαίου να τονιστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. Δεν είναι άλλωστε και μυστικό πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η στρατιωτική ωφέλεια του προγράμματος Γαλιλαίος. Και συχνά προβάλλεται η απέτηση για την επέκταση, αν θέλετε, της χρήσης του Γαλιλαίου σε στρατιωτικές χρήσεις. Ρωτώ λοιπόν, πώς, ε, σε ποιο βαθμό επιτρέπεται τα χρήματα αυτά που χορηγούνται για το Γαλιλαίο να προέρχονται από πολιτικά κονδύλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λόζιν. Κυρία Λόζιν, υπάρχει άλλος ομιλητής που θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις έχω να απευθύνω προς ε, τον επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Κέντρου. Καταρχάς σας ικανοποιεί το στάτους ως ε, εξωτερική υπηρεσία. Κατά δεύτερον, πώς θα επιδράσει στο μέλλον το πρόγραμμα Γαλιλαίο στο πρόγραμμα δράσης σας και κατά τρίτον σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία για το 2005 το 36% ε, αφιερώθηκε για την ειρήνη 15% το 2006, 26% και σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια 17% και μόνο 2% το 2008. Βλέπουμε λοιπόν μια σαφή καθοδική τάση. Υπάρχει κάτι ενδεικτικό σε αυτή τη στάση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καθώς ε, έχουμε μαζί μας πέντε εμπειρογνώμονες για τις απαντήσεις. Θα ήθελα να σας ζητήσω να περιοριστείτε στις απαντήσεις σας σε 5-6 λεπτά, αν γίνεται. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σχετικά με την ερώτηση τη σχετική με την πρόσβαση στις εμπορικές εικόνες, εμπορικές φωτογραφίες από μη ευρωπαϊκές πηγές και σε συνεργασία και για την συνεργασία με τη ΣΥΠΑ, εμείς αγοράζουμε αυτές τις εικόνες από εμπορικές εταιρείες από τις Ηνωμένε Πολιτείε εδώ και αρκετό καιρό και έχουμε μια καλή εμπορική συνεργασία στον τομέα αυτό. Όμως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι μη Ευρωπαίοι παροχή υπηρεσιών. Εξετάζουμε λοιπόν την δυνατότητα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία να είναι εγγυημένα από Ευρωπαίους παροχής. Είναι και οικονομικό το θέμα αλλά μιας και είναι περιορισμένος ο προϋπολογισμός μας, 12,3 εκατομμύρια ευρώ, 9 εκατομμύρια πηγαίνουν ε, στην αγορά των εικόνων και αυτό διαιρείται από 27 σε 27 ε, κράτη-μέλη. Ενώ υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι εδώ που εργάζονται σε υπηρεσίες με μεγαλύτερους προϋπολογισμούς. Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε όμως και την αλλαγή του ορισμού των κοινών δράσεων που καθορίζει το περιβάλλον εργασίας των κέντρων, το οποίο αποφάσισε να διευρύνει τον κατάλογο των τρίτων χωρών με τις οποίες ε, μπορεί να συνεργαστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δορυφόρων ε, ε, και να πει ότι συνεργαζόμαστε όχι μόνο με ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ αλλά με γενικά μέλη του ΝΑΤΟ και αυτό σημαίνει Ηνωμένε Πολιτείες και Καναδάς. Έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα ξεκινήσει με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας του Διαστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζουμε ότι τέτοιου μορφές συνεργασίες, σύνεργασίες στο μέλλον θα αναπτυχθούν σε προγράμματα τα οποία είναι σχετικά με τις ανάγκες που έχει το κέντρο δορυφόρων. Σχετικά τώρα με την ερώτησή σας για το καθεστώς του κέντρου δορυφόρων σαν ανεξάρτητης υπηρεσίας. Θα πρέπει να πούμε ότι η δομή του κέντρου αυτού είχε καθοριστεί το 2001 όταν το κέντρο έγινε τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από το σημερινό. Το κέντρο δορυφόρων μόλις είχε αξίσει, αρχίσει τότε να λειτουργεί και άκουσα ότι είμαστε θύμα της επιτυχίας μας. Όχι, δεν υπάρχουν θύματα ανάμεσά μας, απλά ε, έχουμε πάρα πολλή δουλειά χάρη στην ταχυτάτη ανάπτυξή μας στον τομέα, τον στρατιωτικό αλλά και τον πολιτικό κυρίως. Σκοπεύουμε λοιπόν οι δομές μας να προσαρμοστούν καλύτερα σε αυτή τη μορφή ε, α, και έρχομαι εδώ στην ερώτηση σχετικά με την αλλαγή των αποστολών της ε, υπηρεσίας δορυφόρων. Πριν μερικά χρόνια μας ζητούσαν συγκεκριμένες αποστολές ε, τα κράτη-μέλη και όχι τόσο συνολικότερα υπηρεσίες. Τώρα όμως ουσιαστικά οι συγκεκριμένες αποστολές ε, στόχοι είναι η βασική μας προτεραιότητα και η διαχείριση των κρίσεων, η υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων ελέγχει επιχειρησιακά το κέντρο και μας στέλνει αυτές τις αποστολές σαν, πρώτη, σαν βασική κάθε φορά προτεραιότητα. Και μιας και ο προϋπολογισμός μας δεν έχει αλλάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο από την προτεραιότητα υπαρίθμου 1. Ελέγχουμε λοιπόν να δούμε αν υπάρχουν και άλλες δυνατότητες έτσι ώστε να μην υπάρχει μόνο ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας αλλά και οργανική ανάπτυξη σχετικά με το Γαλιλαίο. Δεν εμπλεκόμεθα στο πρόγραμμα Γαλιλαίο σε αυτή τη φάση, αλλά κάθε εξέλιξη στον τομέα του διαστήματος και της ασφάλειας θα βοηθήσει νομίζω να λαμβάνονται πιο σωστές αποφάσεις στον τομέα τον οποίο εμείς καλύπτουμε. Ευχαριστώ κύριε Φιντά. Θέλετε να δώσετε κι εσείς κυρία Ράης απαντήσεις. Πάρα πολύ σύντομα. Συμπληρώνοντας τις πληροφορίες που έδωσαν οι συνάδελφοι. Έχουμε ένα πολύ σαφές πλαίσιο το οποίο καθορίζεται από το κοινό πρόγραμμα δράσης και οι μόνες χώρες οι οποίες μπορούν να συνδεθούν με τις εργασίες μας είναι οι χώρες που ανήκουν στο ΝΑΤΟ αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υποψήφιες χώρες. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το πώς και πού μπορούν τα προγράμματα αυτά να αναπτυχθούν. Οι χώρες αυτές όμως μπορούν να ζητήσουν συγκεκριμένες αποστολές από το κέντρο και λαμβάνονται οι αποφάσεις ανάλογα αν μια τέτοια αποστολή θεωρείται χρήσιμη για την συζήτηση γύρω από τα θέματα της ΚΕΠΑ και της πολιτικής ασφάλειας ή αν είναι μια αποστολή την οποία ζητά ένα κράτος μέλος, το κράτος μέλος αυτό θα αποφασίσει αν το προϊόν το οποίο έχει ζητήσει θα διανεμηθεί και στις υπόλοιπες χώρες. Να σας θυμίσω εδώ ότι όλα τα προγράμματα, τα προϊόντα μάλλον του κέντρου πηγαίνουν αυτόματα σε όλες τις χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλές φορές συνεργαζόμαστε με διάφορα κράτη-μέλη, χώρες του ΝΑΤΟ πάντα, οι οποίες μπορεί να ζητούν συγκεκριμένες αποστολές και υπηρεσίες από το κέντρο ή μπορούν να αποσπούν υπαλλήλους στο κέντρο. Όπως είπε ο Διευθυντής, οι απαιτήσει τα τελευταία χρόνια έχουν διπλασιαστεί. Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή τη στιγμή μια αποστολή χρησιμοποιεί το κέντρο ε, για τα προϊόντα τα οποία επιθυμεί. Από εκεί και πέρα η χρήση του κέντρου μας αυξάνεται συνεχώς. Έτσι και σε επίπεδο στρατιωτικής ε, αλλά και πολιτικής ε, δραστηριότητας συνεργαζόμαστε πλήρως σε τομείς προβληματικούς όπως η Γεωργία, το Κωσυφοπέδιο, η Ουγγάντα κτλ. για την ερώτηση της κυρίας Γκόμες και για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχω εδώ να δώσω συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το τι αλλαγές υπάρχουν με την κυβέρνηση Ομπάμα. Περιμένουμε την αναθεώρηση της πολιτικής αυτής όταν ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Βέβαια οι σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντικές σε επίπεδο διαλόγου Συνεργαζόμαστε φυσικά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες υπηρεσίες που εκπροσωπούνται εδώ στα πλαίσια του διαλόγου που οργανώνεται στη Ουάσιγκτον γύρω από το διάστημα τους επόμενους μήνες. Πώς τώρα, ή αν κατάλαβα καλά, πώς ε, συνεργαζόμαστε με την ε, ύπατη εκπρόσωπο για τις εξωτερικές σχέσεις και τους άλλους εμπλεκομένους. σε λειτουργικό επίπεδο. Έχουμε τον διαρθρωμένο διάλογο για το διάστημα που βοηθάει ιδιαίτερα. Έχει τις δικές της αρμοδιότητες, η ύπατη εκπρόσωπο σχετικά με τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τις εργασίες μας. Το κέντρο παραμένει κάτω από τον πολιτικό έλεγχο της ΚΕΠΑ, έχει σημασία αυτό. υπάρχει πολιτικός έλεγχος από πλευρά του PSC και θεωρούμε θα υπηρεσία του Συμβουλίου. Αυτά όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν δημιουργείται ε, στη συγκεκριμένη φάση η εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άλλα κέντρα εργάζονται κυρίως για την τεκμηρίωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από πλευρά Συμβουλίου και υπάρχουν θέματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν, όπως είπε η κυρία Γκόμες, σχετικά με τις εξωτερικές δράσεις. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ κύριε Ράις. Ο Ναύαρχος Τριουλέρ. Θα πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι ο κεντρικός τομέας εξυπηρετείται από τις εγκαταστάσεις και από τις υπηρεσίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Βάση Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Δυνατότητας. Θα πρέπει να διαμορφωθούν ορισμένες σχέσεις, οι οποίες τώρα έχουν ξεκινήσει με τις Ηνωμένε Πολιτείε κυρίως, αλλά προς το παρόν όχι, όχι στα διαστημικά θέματα και παραμένουμε πάντα σε ένα πλαίσιο απλής ανταλλαγής πληροφοριών και θεμάτων πάνω στα οποία έχει ξεκινήσει η συζήτηση με τις Ηνωμένε Πολιτείε αφορούν άλλες δυνατότητες όπως τα ελικόπτερα. Πάντως στον τομέα του ελέγχου του διαστήματος είναι ένας τομέας πάρα πολύ ευαίσθητος και δεν μπορούμε παρά να έχουμε στενότερες σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Δεύτερο ερώτημα αφορά τις στρατιωτικές χρήσεις του Γκαλιλαίου. Εδώ είμαστε παρουσία ενός συστήματος το οποίο αναπτύχθηκε πλήρως στα πλαίσια μιας πολιτικής πρόπτικης. Παρ' όλα αυτά οι χρήσεις του Γκαλιλαίου και μία από τις υπηρεσίες που παρέχει το PRS ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον τομέα της άμυνας. Ξεκινήσαμε λοιπόν, και αυτό είναι σχετικά πρόσφατο, μια διαδικασία σύνδεσης και επικοινωνίας με την διοικητική δομή του Γκαλιλαίου για τη στρατιωτική χρήση ορισμένων υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει τον Γκαλιλαίο. Ένα από τα θέματα αφορούσε την συνεργασία της δραστηριότητας διάστημα και ασφάλεια και αν κατάλαβα καλά το ενδιαφέρον της δημιουργίας μιας ξεχωριστής μονάδας. Δεν θα δώσω πολιτική απάντηση γιατί δεν είναι στο επίπεδό μου, αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα που δείχνει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να γεννήσει μορφές συνεργασίας και αναφέρθηκα στον τομέα της, ε, του ελέγχου του διαστήματος εδώ έχουμε ένα υποδειγματικό θα έλεγα πεδίο όπου εξ αρχής ε, οι ανάγκες των πολιτικών χρηστών και των στρατιωτικών χρηστών αναπτύχθηκαν από κοινού με μία μόνιμη συνεργασία και με μόνιμες ανταλλαγές απόψεων καταλήξαμε σε εκπεφρασμένες ανάγκες, διαφορετικές μεν μεταξύ τους, αλλά που έχουν και ένα μεγάλο κοινό τμήμα. Μου φαίνεται λοιπόν ότι πριν αρχίσουμε να συζητάμε για, υπο... για δομές, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε το τι προστιθέμενη αξία προσφέρουν τα ίδια τα προγράμματα όταν εμπλέκουν και πολιτικούς και στρατιωτικούς ε, πρωταγωνιστές αυτά. Ευχαριστώ βάρχε. Η κυρία Χάιντς Κούμπερ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι πολλές ερωτήσεις αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διαστημική δραστηριότητα δεν μπορεί να ειδωθεί απομονωμένα πάντα πρέπει να αναζητούμε μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ του που θα έχουμε αυτονομία για παράδειγμα σε συγκεκριμένους τομείς ασφαλείας όπου πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τις δικές μας δυνατότητες που θα μας παρέχουν ανεξάρτητες πληροφορίες και από την άλλη πλευρά όμως ε, πρέπει να μπορούμε να αξιολογούμε όπου υπάρχουν ανάγκες συνεργασίας με σημαντικούς εταίρους όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία και άλλες χώρες που έχουν πρόσβαση στο διάστημα. Υπάρχουν ε, βεβαίως ε, νομοθεσία που καλύπτει αυτά τα πράγματα σε δομικό πλαίσιο και υπάρχει για παράδειγμα ο διάλογος που έχουμε ξεκινήσει με τις Ηνωμένε Πολιτείες, με τη Ρωσία, με την Νότια Αφρική επίσης ε, και άλλες χώρες που έχουν πάει στο διάστημα Πέρα όμως από αυτά υπάρχουν και άλλα κανάλια, άλλοι διαλόγοι που μας επιτρέπουν να εξετάζουμε τομείς με δυνατότητα συνεργασίας για τις εφαρμογές που έχουν να κάνουν με το διάστημα και τις οποίες αναπτύσσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαν να πούν περισσότερα εδώ οι συνάδελφοι από τον Καλλιλέο, αλλά για παράδειγμα πρέπει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες καθώς αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ενδεχομένως για 80% των απαιτούμενων πληροφοριών για την ασφάλεια στο διάστημα. καθώς αυτά τα στοιχεία προέρχονται προς το παρόν από αμερικανικές πηγές. Χρειάζεται λοιπόν οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με την διεθνή συνεργασία. Ετέθη ένα ερώτημα για την συνθήκη για το εξώτερο διάστημα και για το αν δραστηριοποιούμαστε για την ενημέρωση της συνθήκης. Δεν είμαστε εμείς ειδικοί, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στην ε, θέση του οδηγού προκειμένου να δημιουργηθεί μήνα κώδικα θεοντολογίας προκειμένου να αποφύγουμε τα απορρίμματα στο διάστημα και επίσης να συμμορφωθούμε με μέτρα διαφάνειας όσον αφορά την κυκλοφορία στο διάστημα. Τώρα, αν υπάρχουν και επιπλέον δραστηριότητες, εγώ δεν τις γνωρίζω όσον αφορά τουλάχιστον αυτή τη συνθήκη που πηγάζει από τον ΟΗΕ και θα θεωρούσε ότι οποιοδήποτε σχετική δραστηριότητα θα έπρεπε να ξεκινήσει από τον ΟΗΕ. Μία άλλη ερώτηση που τέθηκε αφορούσε τη χρηματοδότηση των διαφόρων ε, ευρωπαϊκών διαστημικών εφαρμογών, GMES και Galileo δηλαδή. Καταρχάς, η κυρία Λέσσινγκ ε, ρώτησε κάτι πιο γενικό. Αν είναι νόμιμο και δυνατό να υπάρξει χρηματοδότηση κυρίως από γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν τα πολιτικά θέματα. Νομίζω ότι ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή ότι αυτά τα συστήματα ωφελούν το πολιτικό τομέα, τον έλεγχο, την κυκλοφορία κτλ. Και άρα είναι προφανές ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τέτοιου είδους γραμμές. και για το Τζιμίς και για τον Γαλιλαίο οι αποφάσεις ελήφθησαν προκειμένου να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, καλύτερα δεδομένα, καλύτερες εικόνες προκειμένου να εφαρμόσουμε για παράδειγμα τις περιβαλλοντικές μας ε, πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και για να εξυπηρετήσουμε εθνικούς πελάτες. Όμως αυτές οι εικόνες μπορούν παράλληλα να χρησιμοποιηθούν και για λόγους ασφαλείας. Αυτό αναφερόταν στην ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος ότι ναι μεν δηλαδή έχουμε σαφείς πολιτικούς στόχους αλλά μπορούν τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτικούς λόγους. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό για τον Γαλιλαίο αλλά και για το συνολικό κόστος του GMES. Θα σας παραπέμψω στους εμπειρογνώμονες για τον Γαλιλαίο και το GMES εδώ στα έδρανα της Κομισιόν. Μου δίνετε την άδεια να τους δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι, μόλις τώρα με ενημέρωσαν ότι έχουμε υπεύθυνου για τον Καλλιλέο εδώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Όσον αφορά τα προγραμματικά θέματα για το GMAS, το 2008 είχαμε έναν κοινοτικό προϋπολογισμό για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GMES και στα πλαίσια της ΓΔ Μεταφορών και Ενέργειας αρχικά και τώρα στα πλαίσια της ΓΔ Επιχειρήσεων οργανώσαμε τα σχετικά θέματα. Όσον αφορά το πρόγραμμα Ίγνος, το ένα από τα δύο είναι σε επιχειρησιακή φάση από πέρυσι. Έχουμε δηλαδή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα πλοήγησης με βάση την Ευρωπαϊκή Εντολή και όσον αφορά το Γαλιλαίο υπογράψαμε τη σύμβαση για τους δορυφόρους και ελπίζουμε ότι θα βρισκόμαστε σε προεπιχειρησιακό στάδιο το 2014 θα έχουν ξεκινήσει ορισμένες υπηρεσίες, συγκεκριμένα η κυβερνητική υπηρεσία, η Τι θα γίνει στη συνέχεια. Είναι προφανές ότι τα προγράμματα αυτά θα εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται από τους δημόσιους πόρους και άρα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στις ε, επόμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές. 2014-2020 μεταξύ άλλων. Οπότε εμείς προετοιμάζουμε ανακοίνωση για την συνέχεια με το 2013 και για τον αντίκτυπο που θα υπάρξει για τις δημοσιονομικές πρόπτικες. Όσον αφορά τις στρατιωτικές εφαρμογές του Γκαλιλαίου, να πω ότι μία από τις πρώτες υπηρεσίες που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν το 2014 το PRS έχουν δυνατότητες ε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, στις ε, πολιτικές ή στρατιωτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Μάιο θα παρουσιάσουμε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις ε, βασικές αρχές αυτής της υπηρεσίας που θα δείχνει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη-μέλη, τις κυβερνήσεις κτλ. Επίσης ε, θα αναφερθεί και το θέμα του πρόσβασης για τρίτες χώρες καθώς και διάφορα που έχουν να κάνουν με τα τεχνολογικά στοιχεία. Τέλος. Όσον αφορά τις αποστολές ΠΕΣΤ, για παράδειγμα, του Γαλιλαίου, τα πολιτικά δηλαδή, δεν υπάρχει πρόβλημα να χρησιμοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει και κάποια κοινή δράση που θα ρύθμιζε τέτοιου είδους αποστολές ΠΕΣΤ, αλλά αυτό βεβαίως δεν είναι θέμα της Κομισιόν. Αυτές τις κοινέ δράσεις τις αποφασίσουν η Προεδρία και τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει ένα γενικό πλαίσιο που θα αναφέρει τις βασικές γενικές αρχές και δεν θα περνάει τόσο σε πιο συγκεκριμένα θέματα όσον αφορά τη διαχείριση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος ε, Ντάμελ, ευχαριστώ σε ό,τι αφορά την συνεργασία. Θα ακούσατε ότι πριν από κάποια χρόνια κατά την αρχή ε, του προγράμματος Γαλιλαίου είχαμε κάποια θέματα με τις, τις Αμερικανικές αρχές. Δεν καταλάβαινα γιατί ήθελε η Ευρώπη να ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό και πήρε κάποιο καιρό μέχρι ότου μας, μας υποστηρίζουν πλέον και τώρα έχουν ανακοινώσει ότι θα είναι και πελάτες του προγράμματος ε, Γαλιλαίο. Είναι μεγαλύτερο ο προπολογισμό των είπα, από ότι όλοι οι άλλοι φορεί στον τομέα αυτό. Άρα δεν θα ήταν σοφό και φρόνιμο το να μην τους λάβουμε υπόψη για το πρόγραμμα δεστητοποίησης για το διάστημα. Ε, εξ αρχής είχαμε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ και πολλά επιχειρήματα χρησιμοποιήθηκαν. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SSA χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την αύξηση από δικής τους πλευράς του, των κονδυλίων του προγράμματος SSA και επίσης θα γνωρίζετε ότι και ο Καναδάς είναι συνεταιρισμένο μέλος ε, της ΕΙΖΑ. Έχουμε καθημερινές λοιπόν συζητήσεις από πλευράς εξάρτησης ό,τι αφορά τα νομικά ζητήματα. Δεν εξαρτάται αυτό από... Η εξάρτηση έχει να κάνει μόνο με τις ε, διαστημικές ε, πτήσεις. Άρα εξαρτόμαστε από εκτοξεύσεις από την Αμερική και τη Ρωσία σε ό,τι αφορά τις εκτοξεύσεις, γιατί δεν έχουμε σχετικές ε, υπόδομες ε, στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο τραύμα πλέον στη ΣΥΠΑ, γιατί θα τεθεί εκτό λειτουργία το σχετικό σκάφο του, αλλά για μα δεν νομίζω ότι από γεωπολιτική άποψη στην παρούσα φάση παρουσιάζεται οποιοδήποτε πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μα με τη ΣΥΠΑ για το που οδεύει η Κίνα τώρα. Όντως έχει διεξάγει η Κίνα ε, ελέγχους για την καταστροφή δορυφόρων πριν από κάποια χρόνο, χρόνια και αυτό για μας ε, παρουσίασε προβλήματα σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα, αλλά από ό,τι ξέρετε απασχολεί πολλούς μηχανικούς και αναπτύσσει την σχετική τεχνολογία με ηλικιώδη ταχύτητα. Έχει αναπτυχθεί στη ΣΥΠΑ ε, μία πολιτική γιατί υπάρχει ο φόβος ότι η Κίνα θα καταστρέψει τα διαστημικά τους, διαστημικές τους υποδομές. Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι η παρουσία των ήπα εξακολουθεί να είναι καταλητική στο διάστημα. Τώρα, ποιες είναι οι αλλαγέ μετά την, τον πρόεδρο Ομπάμα σε ό,τι αφορά τη διάσταση της ασφάλειας δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Τα βασικά δόγματα των Αμερικανών, όπως για παράδειγμα η ενωτερότητα σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες έχουν παραμείνει τα πράγματα όσα έχουν, αλλά αναζητούνται νέοι στόχοι στον τομέα του διαστήματος. Δεν μπορούν πλέον να ταξιδεύουν στο φεγγάρι, στον Άρη, άρα αναζητούν νέες ε, κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει μια τεράστια ευκαιρία για μας στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη διερευνητική φάση και αυτό αναγκάζει τους Αμερικανούς να συνεργαστούν μαζί μας. Άρα μάλλον θετική είναι η εξέλιξη. Επίσης για την ερώτηση για τη συνθήκη της Λισαβόνας, κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει άλλη ευρωπαϊκή υπηρεσία. Νομίζω ότι έχει καταδείξει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο πόσο ικανή είναι και να δεν θα πρέπει να δημιουργούνται αλληλεπικαλύψει. Αυτά, πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πολύ. Λέει ο πρόεδρο, να ευχαριστήσω και όλου του εμπειρογνώμονες εξ ονόματο τη Επιτροπής μα, τη Υποεπιτροπής μας. Είμαι βέβαιο ότι έχουμε ενημερωθεί πολύ καλύτερα πλέον και είμαι βέβαιο ότι πρόκειται για μια πρώτη συνάντηση, όχι όμω για την τελευταία συνάντηση στα πλαίσια τη Τρέχουσα Νομοθετική θητεία. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να κάνουμε ένα και δύο λεπτών για να δώσουμε και την ευκαιρία στους ε, καλεσμένους μας που πρέπει να φύγουν να αποχωρήσουν και θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο τμήμα της ε, ακρόασής μας σε λίγα λεπτά με τον πρόεδρο Μαυρονικόλα. Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε το δεύτερο τμήμα της ακρόασης. Please get your seats. Ευχαριστούμε. Το δεύτερο τμήμα θα είναι για την έρευνα για την ασφάλεια και έχουμε μαζί μας τον κύριο Κρίστιαν Μπρέαντ, Διευθυντή Έρευνας και Τεχνολογίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Και τον κύριο Κρίστοφ Κάουτσου υποδιευθυντή τη Μονάδα Έρευνας και Ανάπτυξης του τομέα της ασφάλειας. Να δώσουμε το λόγο στους δύο μιλητές. Αν θα μπορούσατε παρακαλώ, παρακαλώ να περιστείτε σε 15 λεπτά για να έχουμε χρόνο και για τις ερωτήσεις μετά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέαντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το έργο της ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ε, και βεβαίως ε, σε σχέση με το θέμα της σημερινής παρουσίασης δηλαδή της ε, έρευνας στον τομέα της ασφάλειας, που στόχος της είναι να καλύπτει τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της Ευρωπαϊκής Άμυνας, κάτι πολύ σημαντικό γιατί διαπιστώνουμε ότι όντως βρισκόμαστε σε δρόμο να καλύψουμε τις ανάγκες των κρατών μελών. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να επενδύουμε σε όλους τους τομείς μεν, αλλά και να επικεντρωνόμαστε σε τομείς που χρειάζονται μεγάλη συνεργασία. Και ο οργανισμός μας συντονίζει διάφορα προγράμματα έρευνας ε, εκ μέρους των κρατών μελών στα διάφορα εργαστήρια των κρατών μελών. Επίσης προσπαθούμε να μειώσουμε την εξάρτηση από βασικές τεχνολογίες κρίσιμας σημασίας. Το θέμα αναφέρθηκε και πριν. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ορισμένες ε, διαστημικές υπηρεσίες που είναι πολύ σημαντικές και πολιτικά και στρατιωτικά και γι' αυτό πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται σε θέση που θα της δίνει τη δυνατότητα πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες σε κάθε περίπτωση. Επίσης προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ε, ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης που συμπεριλαμβάνει και τα ερευνητικά κέντρα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τέλος προσπαθούμε να αυξήσουμε τις συνέργειες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Βλέπετε εδώ κάποια διαγράμματα για να δείτε ποιες είναι οι επενδύσεις για την τεχνολογία άμυνας από το 200 δις συνολικά, 2,5 δις αφορούν την άμυνα και έχουμε μια μικρή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε αρκετά μεγάλη συνεργασία κρατών μελών για ποσό που αφορά περίπου 400 εκατομμύρια. Επίσης να πω ότι σε αντίθεση με άλλους τομείς αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μεγάλη συμμετοχή των κρατών μελών, ειδικά Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας, ενώ ακολουθούν Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, κατοχώρες και Σουηδία που αφορούν ένα 33% ενώ οι υπόλοιπες χώρες ε, εκπροσωπούν μόνο το 1% με την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να μοιράζονται το 64% των επενδύσεων. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε κάνει αρκετά συνεργασίες. Μπορείτε να δείτε εδώ στοιχεία για τα τρία τελευταία χρόνια και βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στη χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Καλό σημάδι αυτό, καθώς αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τον προϋπολογισμό ενώ παράλληλα τα κράτη-μέλη, αρκετά κράτη-μέλη θεωρούν ότι πρέπει να αυξηθεί η συνεργασία και εφόσον μειώνεται ο προϋπολογισμός καταλαβαίνουν ότι πρέπει να μοιραστούν και αυτοί τους πόρους τους προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτούς τους νέους εξοπλισμούς. Ορισμένα παραδείγματα προγραμμάτων για τα οποία θα επενδύσουμε πολλά τα επόμενα χρόνια. MMCM. Θαλάσσια μέτρα καταπολέμησης ναρκών. Είχαμε καλή συνεργασία φέτος και μάλλον θα ξεκινήσει το επόμενο έτος. Μετά το CBRN, στο οποίο θα αναφερθώ και στο δεύτερο τμήμα της ομιλίας μου. και τρίτο πρόγραμμα Counter IED όπως γνωρίζετε πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό καθώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα στρατιωτικά μήματα. Περνάω τώρα στην ε, πρωτοβουλία συνεργασίας ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκίνησε πέρυσι και επίσης με την ΕΣΑ και την ADA. Προσπαθούμε να συγχρονίσουμε τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Υπηρεσίας Διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε πιο συστηματική τη συνεργασία και ελπίζουμε ότι με το 7 πρόγραμμα πλαίσιο θα μπορέσουμε να καταφέρουμε ακόμη περισσότερα όσον αφορά την ανάπτυξη εργαλείων για την ασφάλεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων. Επαναλαμβάνω, το βασικό είναι να έχουμε συγχρονισμό των δραστηριοτήτων και μεγιστοποίηση των συνεργειών. Και βεβαίως θα λαμβάνουμε συνενετικές αποφάσεις προσπαθώντας να βελτιώσουμε την εφαρμογή. Είχαμε μία συνάντηση με την ΕΖΑ πρόσφατα και έχουμε ήδη εντοπίσει κάποιους πολλά υποσχόμενους υποψήφιους όπως το CBRN, το UAS καθ όπου μας ενδιαφέρουν και τα υπτάμενα συστήματα αλλά και η διερεύνηση των συστημάτων ενώ ένα τρίτο υποψήφιο πρόγραμμα αφορά την γνώση των καταστάσεων με θέματα όπως οι αισθητήρε, η κυβερνοασφάλεια και η διαχείριση πληροφοριών. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα υπάρξει αυξημένη τάση στο μέλλον για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Τελειώνοντας και προκειμένου να προλάβω κάποιες ερωτήσεις από το κοινό, να σας αναφέρω και τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει η συνθήκη της Λισαβόνας όπως γνωρίζετε στο άρθρο 179 συνθήκες της Λισαβόνας αναφέρεται ότι θα είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενίσχυση της ε, τεχνολογικής βάσης προωθώντας όλες τις σχετικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις συνθήκες. Επίσης αναφέρεται ότι όλες οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων επίδειξης θα αποφασίζονται με βάση τις διατάξεις αυτού του τίτλου. Άρα υπάρχει αναφορά όχι μόνο στο άρθρο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας αλλά και στο άρθρο 179, κάτι που διαφοροποιεί πολύ την κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν. Και βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ένα από τα κύρια μέρη μαζί με το Συμβούλιο όπου θα ληφθούν αυτές οι αποφάσεις. Και βεβαίως ε, μας επιτρέπουν να κάνουμε και έρευνα με βάση το ανθρώπινο δυναμικό με χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ε, και να γνωρίζουμε ότι σύντομα θα χρειαστεί να απαντηθούν τέτοιου είδους ερωτήματα. Αυτά από εμένα και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριο Σκάουτς. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση. Θα πρέπει δυστυχώς να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του κυρίου Μαλακάρνε, ο οποίος βρίσκεται σε συνάντηση με τον Επιτρόπο Ταγιάννη. Καταρχάς, να εξηγήσω που βρισκόμαστε σήμερα σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας στο πρόγραμμα πλαίσιο, ε, το πέμπτο λοιπόν, ορισμός ε, ξεκίνησε από το 2002-2003 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε πάρα πολύ δραστηρία για την διατύπωση της ομάδας των προσωπικότητων ε, που έφερε αν θέλετε μαζί βασικούς εμπλεκόμενους φορείς ε, για να διαμορφωθεί η μορφή της πολιτικής και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει προσανατολισμός στην έρευνα ε, στην αποστολή, στις συγκεκριμένες αποστολές, όχι γενικά στην έρευνα. Οι συζητήσεις ε, έλαβαν υπόψη του τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον τομέα της έρευνας. Αυτό δεν ε, ήταν εύκολο να απαντηθεί στα πλαίσια της συνθήκης της Νίκαιας. Και τότε βρήκαμε τον εξή συμβιβασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτεί έρευνα σε ό,τι αφορά θέματα ιστορικής ασφάλειας πρωτίστως αυτό και υπό το φως ε, της ε, προσπάθειας που γινόταν τότε για την αστυνομική συνεργασία. Ξεκίνησαν ε, προπαρασκευαστικές εργασίες σε ύψος 15 εκατομμυρίων ευρώ και με την ε, μεγάλη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 7ο στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έδωσαν ε, μια ξεχωριστή διάσταση στο θέμα αυτό με προπολογισμό των 4,5 δισεκατομμύρια στην περίοδο 2007-2014. Καταρχάς να υποστηριχθούν, ο σκοπός ήταν να υποστηριχθούν οι διαδικασίες και οι πολιτικές σε ό,τι αφορά την, τον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, αλλά και σε ό,τι αφορά την ενέργεια και την ασφάλεια. Και σκοπός είναι να πληρωθούν τα χάσματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις υποδομές μέσω τώρα στην Επιτροπή έχουμε 300 εκατομμύρια ε, ευρώ για 80 περίπου project και αν ε, καταμετρήσουμε πόσοι φορείς εμπλέκονται. Είναι λίγο πολύ 800 στον αριθμό περίπου. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα project είναι ευρύτατα στο φάσμα τους από προστασία υποδομών ως ε, προγράμματα διαχείρισης κρίσεων αλλά και πιο πανεπιστημιακά προγράμματα όπως ε, προγράμματα πρόβλεψης για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε κάποια προγράμματα, προγράμματα σε ό,τι αφορά την, ε, τα ναυτιλιακά σύνορα. Και ξεκίνησε μόλις ε, ένα σχετικό project ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ που σκοπό έχουν να τεθούν τα τεχνολογικά α, θεμέλια για τον ε, έλεγχο των ναυτιλιακών συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ανάλογα και με τις ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, για παράδειγμα, ε, ένας τομέας είναι ο τομέας της πολιτικής προστασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Κατά δεύτερον, προστασία ε, των υποδομών, όπου εξετάζουμε τις ενεργειακές υποδομές, τις υποδομές ICT και το καθεξής και έχουμε και το θέμα και της συνοριακής ασφάλειας και σας ανέφερα μόλις το σχετικό παράδειγμα. Έχουμε και το θέμα, το τομέα, τον κλάδο της ε, διαχείρισης κρίσεων. Έχουμε τον τομέα της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, των ε, επικοινωνιών και το καθεξής. Έχουμε τον τομέα της ασφάλειας στην κοινωνία, γιατί οτιδήποτε άπτεται της πολιτικής ε, ασφάλειας αποτελεί κρίσιμο θέμα ασφαλώς. Και έχουμε επίσης και τον τομέα της ε, ευρωπαϊκής έρευνας. Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν σήμερα. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον. Θα βασιστώ σε κάποια έγγραφα τα οποία πρόσφατα δημοσίευσε είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε το άστρεφ το οποίο θα το αναφέρω και σε λίγο πάλι ο πρόεδρος Μπαρόσο στις κατευθυντήριες γραμμές τόνισε την πτυχή της εξωτερικής ασφάλειας και είπε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητές μας για να καταστούμε μια δύναμη πολιτική για την οικοδόμηση και την διατήρηση της ειρήνης. Προσφάτως, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων ε, ενέκρινε μία στρατηγική η οποία έθεσε το σύνδεσμο αυτό μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας και είπε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ιστορική ασφάλεια χωρίς την εξωτερική διάσταση, γιατί η, εσωτερική ασφάλεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την εξωτερική ασφάλεια. Επειδή δύο έχουμε ένα φόρουμ το οποίο εξετάζει το μέλλον της ε, ευρωπαϊκής έρευνας με, χρονική, ε, με χρονικό ορίζοντα το 2015-2020. Η ομάδα αυτή δεν ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά συμμετείχε σε αυτή την ομάδα όλα τα κράτη-μέλη, ο κλάδος, τα πανεπιστήμια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κυβερνητικέ οργανώσεις και υπογραμμίστηκε ότι είναι όλο και πιο σημαντικό να εξεταστεί η εξωτερική διάσταση και αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν προγράμματα υποστήριξης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων. Υπήρξε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2007, το Δεκέμβριο, όπου και αναφέραμε την αρχική μας τοποθέτηση για την έκθεση της πλατφόρμας αυτής και αναφέραμε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί ο τομέα ε, και σε ό,τι αφορά την προστασία των πολιτών. Είπαμε λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον αυτών των κλάδων. Η συνθήκη τη Λισαβόνα, την οποία ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής, όντως αναφέρει ότι η έρευνα μπορεί να καλύπτει όλα τα κεφάλαια όλων των συνθήκων για τη λειτουργία της Ένωσης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει μια σειρά καθηκόντων τα καθήκοντα του Πίτερσμπουργκ, όπως αναφέρεται. σε ό,τι αφορά ανθρωπιστικούς στόχους για την διαχείριση των κρίσεων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ούτω καθεξής. Να περάσω τώρα στα στοιχεία που ανέφερε και ο συνάδελφος ε, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Μπορεί η συνθήκη της Λισαβόνας να επιτρέπει την έρευνα για την άμυνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να κάνουμε την έρευνα αυτή. Στην παρούσα φάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε ακόμα μορφωμένη άποψη. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι πρόκειται για ένα πολιτικό, άκρος πολιτικό θέμα. Να διεξαχθεί σχετική έρευνα. Αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε τι πιστεύουν και οι εμπλικόμενοι φορεί. και σαφέστατα να ακούσουμε τι πιστεύει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρα από την έρευνα για την άμυνα, να δούμε πού συνεργαζόμαστε ήδη με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα στην ε, τεχνολογία με τη χρήση εργαλείων και στο σχετικό συγχρονισμό στον κλάδο αυτό. Ο κύριος Μπρεάντ σας ανέφερε τι ε, πραγματοποιείται, τι εκτελείται στους τομείς αυτούς. Να υπογραμμίζω τα εξής δύο στοιχεία. Είναι καλό να εξετάζουμε μορφές συνεργασίας σε ό,τι αφορά τις tool-based τεχνολογίες, βάσει εργαλείων δηλαδή, υπό δύο όρους, ότι θα πρέπει να υπάρχει καταρχάς όφελος, δεν ε, θα πρέπει να πρόκειται για αδιέξοδα και Δεύτερος όρος, ότι δεν θα πρέπει να παραμελούμε το σκέλος, ε, την διάσταση της κοινωνίας και τι εννοώ ο αντίκτυπος ε, σε ό,τι αφορά τα ήθη κτλ. δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές χρήσεις αλλά όταν πρόκειται για θέματα πολιτικής ασφάλειας και έρευνας πολιτικής ασφάλειας είναι πολύ μεγαλύτερος ο σχετικός αντίκτυπος και στο σημείο αυτό θα ήθελα να κλείσω την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις τώρα. Κοπά. Κύριε Κοπά. Uh, uh, να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές για την παρουσίασή τους. Όντως, η έρευνα στον τομέα της ασφάλειας είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ τον δεύτερο ομιλήτη το εξής. Άκουσα με ενδιαφέρον Του τομείς προγραμμάτων με τα οποία ασχολείστε. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος ορίζει την προτεραιότητα με την οποία εφαρμόζονται τα προγράμματα και πώς ακριβώς ε, γίνεται η συνεργασία, πώς λειτουργεί η δομή. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι είμαστε ακόμη στις αρχές, αλλά θα με ενδιαφέρε πολύ να ακούσω πώς λειτουργεί το σύστημα. Σα Σας ευχαριστώ. Σε σχέση με αυτά που παλιά άκουγα όταν ήμουν νέα, και αυτά που μάθαινα, όπου η ασφάλεια και η άμυνα πάντα είχαν να κάνουν με εξωτερική επίθεση. Η άμυνα ήταν κατά μία εξωτερική επίθεση. Σε σχέση λοιπόν με αυτά που μάθανα παλιά, έχει αλλάξει πάρα πολύ η έννοια της ε, επίθεσης και της άμυνας. Αυτά που μας παρουσιάζεται είναι πόσο έντονη είναι η σχέση μεταξύ ιστορικής και εξωτερικής ασφάλειας σήμερα και νομίζω ότι επειδή πραγματικά είναι έντονη αυτή η σύνδεση και αυτή η σχέση, έχουμε μεγάλες ανάγκες για διαφάνεια και δημοκρατία στον τομέα αυτό. αναφέρθηκε κάμποσες φορές στο πρόγραμμα ΕΣΡΕΦ. Και κάποιες από τις συστάσεις αυτές ε, πρέπει να σας πω ότι τι εξέτασα πριν από την συνάντηση αυτή και κάποιες ε, συστάσεις έχουν να κάνουν με τα προγράμματα έρευνας και ανακύπτει κάπως η σκέψη, η υποψία ότι μιλάμε για την ασφάλεια των πολιτών αλλά αναφέρεται για παράδειγμα η αντιμετώπιση πολιτικών ε, κινημάτων, πολιτικών ε, κινημάτων ριζοσπαστικοποίησης και το καθεξής. Νομίζω λοιπόν ότι το πρόγραμμα αυτό έχει να κάνει και με το κράτος και με τη διαμόρφωση, τη μορφή του κράτους. Το φόρουμ λοιπόν αυτό συμπεριλαμβάνει διάφορους ε, τομείς ε, της κοινωνίας των πολιτών. Νομίζω ότι δεν είναι αρκετή η συμμετοχή όμως της κοινωνίας των πολιτών. Και κοιτώντας πόσο επηρεάζει η έρευνα αυτή και ιδιαίτερα πόσο θα επηρεάσει στο μέλλον ο αντίκτυπος της έρευνας, κατά την εφαρμογή της δηλαδή, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποια η τοποθέτησή σας για την πιο έντονη συμμετοχή στην διαδικασία αυτή των ε, ενώσεων για παράδειγμα ε, πολιτικών δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικτύου για την ειρήνη και διαφόρων άλλων τέτοιων οργανώσεων και ενώσεων. Γιατί θεωρώ ότι είναι έντονη η υποεκπροσώπηση των τομέων αυτών. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση από την πλευρά των απλών Ευρωπαίων πολιτών που χρηματοδοτούν αυτά τα προγράμματα έρευνας για τον τομέα της ασφάλειας είχαν ξεκινήσει το 2002-2003 και μέχρι σήμερα περίπου 300 εκατομμύρια έχουν επενδυθεί σε περίπου 80 προγράμματα. Δεν αμφιβάλλω ότι τα περισσότερα από αυτά είναι χρήσιμα και ότι βεβαίως η έρευνα σε τέτοιους τομείς ε, κάποτε έχει θετικά αποτελέσματα, κάποτε όχι. Συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της ασφάλειας των συνόρων. Όμως, πρόσφατα είχαμε συζητήσει σε μια ακρόαση εδώ στην Επιτροπή για το πρόγραμμα Αταλάντα στον Ινδικό ωκεανό. στα παράλια του κέρατος της Αφρικής και είχε αυξηθεί η εφαρμογή, είχαν ε, σταματήσει 11 πλοία Αυτά για το Αταλάντα. Για τα υπόλοιπα 80 προγράμματα και τα περίπου 300 εκατομμύρια έχετε να μας δείξετε άλλα απτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις. Κύριε Μπρέαν, έχετε το λόγο για απαντήσεις. Ε, on uh, question uh, were... Για τις διάφορες ερωτήσεις να πω ότι όταν μιλάμε για την προτεραιοποίηση των προγραμμάτων, οι επιλογές γίνονται από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά που αποφασίζουν πού θα επενδύσουν και ανάλογα θα επιλέξουν τους εξοπλισμούς και εμείς είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. σχετικά με τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας στις εξωτερικές σχέσεις. Αν πάρει κανείς το παράδειγμα του Αφγανιστάν, όπου έχουμε στρατό αυτή τη φάση, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν σαν τελικό στόχο να βελτιώσουν τις συνθήκες εσωτερικής ασφαλείας. Αυτός είναι ο κυρίαρχος στόχος. Και αυτό επιδιώκουμε με αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις. σχετικά με το τι δυνατότητες δίνει επιπλέον η συνθήκη της Λισαβόνα στον τομέα της έρευνας. Ζητήθηκε να παράγουμε για το Υπουργείο Άμυνα στο δικό μας κάποια στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω των νέων προβλέψεων μπορούμε να σας ενημερώσουμε για το περιεχόμενο αυτής της προσπάθειας, αυτής της εργασίας. Αν συγκρίνουμε αυτά με ό,τι είπε ο Κρίστοφ για τα συμπεράσματα της ομάδας των εμπειρογνωμόνων όταν ξεκίνησαν τα προγράμματα ασφαλείας στο τέλος του 2008, Προφανώς το λιτοτερικό του Υπουργείου Άμυνα αναπτύσσοντας στρατηγικές που καλύπτουν τις ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου. Ξέρουμε τι δυνατότητες έχουμε και τι βελτιωμένες ευκαιρίες έχουμε στον τομέα της έρευνας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ασφάλεια. Συμφωνώ με τον Κριστόφ ότι οι αποφάσεις στον κλάδο αυτό είναι πολιτικές αποφάσεις από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Είμαστε εδώ όμως για να βοηθήσουμε, να προσφέρουμε ιδέες και να αναφερθούμε στις δυσκολίες και τις απειλές τις οποίες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Κάουτς. Για την πρώτη ερώτηση, για το πώς θα καθορίσουμε τις προτεραιότητες των προγραμμάτων μας στο εσωτερικό της ομάδας των εμπειρογνωμόνων υπήρχε μια εσωτερική ομάδα, η συμβουλευτική ομάδα για την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας. Είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί αρκετά χρόνια και καθόρισε τους τεχνολογικούς τομείς όπου το πλαίσιο, το έβδομο πλαίσιο θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο. Πήραμε τα αποτελέσματα αυτής ε, της ομάδας, συμπεράσματα αυτής της ομάδας, σαν κατευθυντήρια γραμμή για τα προγράμματα που θα ακολουθήσουμε. Σε οργανωτικό επίπεδο αυτό. Προσπαθήσαμε να καθορίσουμε τις προτεραιότητές μας σε συνεργασία και με τις άλλες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα αποτελέσματα Σε τεχνικό επίπεδο προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τα προγράμματα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα πρώτα να είναι προγράμματα στραμμένα προς τη βελτίωση της ε, τεχνολογίας και μετά από αυτά προγράμματα τα οποία να ενσωματώνουν τα προϊόντα αυτών των τεχνολογιών και να δημιουργούν συστήματα και υποσυστήματα. για το πώς συνεργαζόμαστε με την υπηρεσία της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Η αλήθεια είναι ότι έχει αναλάβει τις υπηρεσίες της, ε, την υπηρεσία της συγγνώμη, εδώ και λίγους μήνες, αλλά συνεργαζόμαστε με τη ΡΕΛΕΞ, τη Γενική Διεύθυνση ΡΕΛΕΞ, που θα είναι τμήμα από εδώ και πέρα ε, της εξωτερικής υπηρεσίας, οπότε έχουμε επαφές. Έρχομαι λίγο στα σχόλια Είπατε ότι έχει αλλάξει ε, η αντίληψη της ασφάλειας ε, και αυτή η σχέση ιστορικής και εξωτερικής ασφάλειας θέτει νέες ε, απαιτήσει ως προς τη δημοκρατία και την διαφάνεια. Συμφωνώ απόλυτα με την εκτίμηση αυτή. Είπατε επίσης ότι στην ΕΣΡΑΦ θα πρέπει να Γίνεται, φαίνεται να γίνονται πιο πολλές προσπάθειες, όχι για τον πολίτη, αλλά πριν από τον πολίτη. Δεν συμφωνώ απόλυτα όμω, ξέρετε, γιατί στο ΕΣΡΑΦ, ξέρετε, υπήρξε μια ομάδα εργασία η οποία ασχολήθηκε αποκλειστικά με το θέμα της ασφάλειας Και τι σημαίνει αυτό σε ό,τι αφορά την διντολογία, την κοινωνιολογία και ούτω καθεξής. Και υπήρξε και στο ΕΣΡΕΦ επίσης μια οριζόντια η ομάδα η οποία προσπάθησε όλα αυτές τις κοινωνικές πτυχές να την περάσει σε όλους τους τομείς εργασίας της ΕΣΡΑΦ και κοιτώντας τα βασικά μηνύματα κλειδί, κλειδιά τα πρώτα τρία μηνύματα έχουν να κάνουν όλα με την κοινωνική πτυχή της ασφάλειας Society and Security, Society and Resilience κτλ αν κοιτάξετε ποιες είναι οι τρεις πρώτες, ε, τα τρία πρώτα μηνύματα, σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών στην ΕΣΡΙΦ. Πάντα θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρειάζεται πιο έντονη συμμετοχή. Αναφέρατε ε, ιδιαίτερα θέματα κρατικής ε, του State Watch μάλλον τις προσκαλέσαμε, αλλά δεν ήρθαν. Σε μία ομάδα εργασία τις προσκαλέσαμε. Αλλά γενικά συμφωνώ μαζί σας ότι τίθενται τεράστιες απαιτήσει ως προς τη δημοκρατία και τη διαφάνεια και σκοπεύουμε φέτος ακόμη να διοργανώσουμε ένα εργαστήρι με το θέμα της ηθικής διάστασης της έρευνας ασφάλειας όπου ακριβώς θα συζητήσουμε τέτοιες ιδεολογικές πτυχές. Στην ανακοίνωση του Δεκεμβρίου του 2009, όπου απαντήσαμε σε θέματα για την ΕΣΡΙΦ, ένα από τα βασικά κεφάλαια πραγματεύεται ακριβώς και αυτή την διεντολογική διάσταση της έρευνας ασφάλειας. Στη συνέχεια ακούσαμε μία ερώτηση για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των έργων μας, των ε, προγραμμάτων μας. Να αναφέρω στο σημείο αυτό ότι ουσιαστικά όλα τα έργα μας, όλα τα προγράμματα που τρέχουν στην παρούσα φάση δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, γιατί τα περισσότερα εξ αυτών οι συμβάσεις ε, οι σχετικές υπογράφησαν τέλη 2008, αρχές 2009, άρα βρίσκονται ακόμα υπό εξέλιξη. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, κάνουμε μία ενδιάμεση αναθεώρηση. Ξεκινάμε μία ενδιάμεση αναθεώρηση για να δούμε τι ακριβώς πέτυχαν τα έργα αυτά, τα προγράμματα αυτά. Μόλις ξεκίνησε αυτή η αναθεώρηση, μόλις έχουμε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, με χαρά μας να σας το διαβιβάσουμε. Μία άλλη παρατήρηση τώρα για αυτά που μας είπε ο Κριστιαν Μπρεάντ. Είπε κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει προσκευαρασκευαστική δράση για την ε, έρευνα αυτή. Δεν είναι ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτής, αυτό ήταν ιδέα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει προπαρασκευαστική φάση για την έρευνα ασφάλειας. Στην παρούσα φάση θα ήθελα απλά να πω ότι εμείς δεν έχουμε διαμορφώσει άποψη, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και συνετοί θεωρούμε και θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό πραγματικά όταν έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας, τον κύριο Μπρεάν, τον κύριο Κότ και ελπίζουμε να σας έχουμε μαζί μας και σε μια μελλοντική συνάντηση. Κλείνουμε στο σημείο αυτό. Θα ξανασυναντηθούμε 26 Απριλίου